Συνάδελφοι, να αρχίσουμε την συνεδρίασή μα. Ελπίζουμε να φτάσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να βρουν τον δρόμο. Έχετε μπροστά σα την ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν έχουμε αντιρρήσει Όχι. Να περνάμε λοιπόν στην έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεων τη 1 η έω 2 Δεκεμβρίου. Κοιτάξτε αν θέλετε τα πρακτικά. Αν δεν μου πείτε τίποτα μέχρι το βράδυ, Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αστάθεις. Έχετε κάτι να μα παρατηρήσετε για τα πρακτικά. Για τα ισπανικά. Ακούγεται ισπανική διερμηνία, λέει η πρόεδρο. Δεν είπα και πολλά σημαντικά, λέει η πρόεδρος. Και περνάμε στι ανακοινώσει του Προέδρου. Αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται στο ίντερνετ και περνάμε στα γερμανικά. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, όχι στα αισθανικά, στα μαλτέζικα, στα αισθανικά, στα σουηδικά. Στις υπόλοιπες γλώσσες έχουμε διερμηνία από και προς. Πάμε στο 4 της ημερήσιας διάταξης για την εκμάθηση κατά την εμπιακή ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Είναι εδώ η εισηγήτρια, η κυρία Χάνιβαλ, θα μας παρουσιάσει το θέμα σήμερα. 14 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Στις 12 το μεσημέρι, 14 Φεβρουαρίου και θα την ψηφίσουμε στις 17 Μαρτίου. Κυρία Χάνιμπαλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πράγματι που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση, ιδίω διότι θεωρώ ότι το θέμα είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε εδώ στην Επιτροπή μας, τουλάχιστον από τότε που είμαι εγώ στην Επιτροπή, το θέμα της ε, παιδείας σε πολύ νεαρή ηλικία. Διότι είναι πολύ σημαντικό ε, ό,τι συμβαίνει με τα παιδιά στην ε, πρώιμη ηλικία τους ε, καθορίζει και τη ζωή τους αργότερα και αν επιλύσουμε προβλήματα θα αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον και επίσης τα παιδιά ε, τα οποία διδάσκονται καλύτερα, μαθαίνουν ε, πολύ καλύτερα και επιτυγχάνουν καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Ε, χαίρομαι λοιπόν που συζητάμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Δεν υπάρχει και μεγάλη έρευνα βέβαια στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και θα σταθώ στην έρευνα σε αγγλόφωνες χώρες, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, και αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει και πόσο επίκαιρο είναι το γεγονός ότι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Από τι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν διαπιστώνουμε ότι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβαση, κυρίω αυτά τα οποία στοχεύουν σε ε, πιο ευάλωτα παιδιά, μπορεί να έχουν σημαντικέ σημαντικές κοινωνικο-οικονομικέ συνέπειες και αυτό συνεχίζεται μέχρι την ενηλικίασή του και στην ενήλικη ζωή του. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο σχολείο, καλύτερου βαθμού, καλύτερε προοπτικέ απασχόληση. Ε, ε, καλύτερη αποζημίωση στην εργασία, λιγότερο έγκλημα, καλύτερη υγεία, καλύτερη οικογενειακή ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ καλά τα πρώτα χρόνια ενό παιδιού και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό για να μπορέσουμε να μην έχουμε μειονεκτήματα σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και να υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα παρακολουθούνται και από διάφορες άλλες παρεμβάσεις όπως υποστήριξη για την εκμάθηση γλωσσών και άλλα θέματα. Μιλάμε λοιπόν για την πρώτη παιδική ηλικία και αυτό το οποίο έχουμε τα πρώτα χρόνια θα συνεχιστεί. Δεν είναι μόνο για τα πρώτα χρόνια, πρέπει να το υποστηρίξουμε και αργότερα και θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο και σε ε, σχέση με την έκθεση. Δυστυχώς σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχουν επενδύσεις για την πρώτη παιδική ηλικία και αυτό σημαίνει ότι είχαμε, έχουμε υψηλότερο επίπεδο δαπανών ε, αργότερα, ε, γεγονός που δεν είναι τόσο αποτελεσματικός προς το κόστος και δεν έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα όσο θα είχαμε αν είχαμε διαπιστώσει το πρόβλημα εξ αρχής. Και επίσης όταν δεν υπάρχουν κατάλληλη ε, παροχή στα πρώτα χρόνια μπορεί να έχουμε και εγκληματικές συμπεριφορές και άλλα κοινωνικά προβλήματα στο μέλλον. Δεν λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ενιαία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ε, παιδεία στα πρώτα χρόνια. Αυτό δεν είναι δυνατόν διότι η Ευρώπη έχει μια ποικιλομορφία πολιτιστικών και εκπαιδευτικών παραδόσεων και ε, η παιδεία στα πρώτα χρόνια παρέχεται με τελείως διαφορετικό τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξει κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζουμε είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ε, αυτή την παιδεία στα πρώτα χρόνια, πώς μπορεί να γίνει καλύτερη και πώς μπορεί να αναγνωρίζεται ακόμα περισσότερο. Επίσης, Υπάρχει και διαφοροποίηση στα κράτη-μέλη ε, ως προς την ποιότητα και παροχή της νηπιακής αυτής παιδείας, πώς παρέχονται υπηρεσίες, πώς ε, διεξάγονται αυτές οι υπηρεσίες. Υπάρχουν ε, τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση λοιπόν διαπιστώνει ότι μία ενιαία προσέγγιση για την ε, νηπιακή ε, εκμάθηση και φροντίδα, την οποία από εδώ και πέρα θα αποκαλώ EC, e η προσέγγιση λοιπόν σε αυτές τις ε, ε, υπηρεσίες ε, δεν μπορεί να είναι ενιαία και θα είναι πολύ δύσκολο και να την υλοποιήσουμε. Θα πρέπει καλύτερα να σταθούμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο θα έχει κοινέ αξίες και στόχους και θα έχουμε ίσως και κάποιες κοινέ δομές. θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να μπορέσουμε να έχουμε παροχή τέτοιων υπηρεσιών και για να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε, καλό θα ήταν να επιτύχουμε ε, ε, να έχουμε καλούς ορισμούς. Νηπιακή ηλικία εννοούμε την ηλικία από 0 έως 6 ετών. Ε, υπάρχουν χώρες στις οποίες ξεκινούν, ξεκινάει η παιδεία πριν από τα 6 χρόνια και φυσικά θα πρέπει να γίνει και κάτι έξω αυτού. Εμείς το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι η μόνη αναφορά που θα κάνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχε μια νομοθεσία για το ε, νηπιακή παιδεία και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και για άλλα κράτη-μέλη. Τα παιδιά στην νηπιακή ηλικία ε, την χάνουν τις μικρότερες δυνατή προσοχής και ε, δαπανώνται και τα λιγότερα. Για την ηλικία από 0 έως 3 ετών ε, δεν υπάρχει καμία σχεδόν φροντίδα και μεταξύ 3 και 6 ετών δεν δίνεται κατάλληλη έμφαση στα θέματα διατροφής και κοινωνικο-οικονομικών ε, ε, παραγόντων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την ε, νηπιακή φροντίδα όχι ως ένα χώρο στον οποίο παρκάρουν οι γυναίκες τα παιδιά τους όταν πηγαίνουν στη δουλειά. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να πηγαίνουν οι γυναίκες στη δουλειά τους, αλλά θα πρέπει οι υπηρεσίες αυτές να μην είναι απλώς ένας χώρος στον οποίο ε, προσέχει κάποιο τα παιδιά και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και πόσο ζωτική σημασία είναι για τα παιδιά να ε, αναπτυχθούν και να μάθουν τα κατάλληλα πράγματα για την ανάπτυξή τους αργότερα. Ιδίω για τα πιο ευάλωτα παιδιά μπορούμε να έχουμε πολύ ε, σημαντικά ωφέλη για το μέλλον και αυτό θα πρέπει να είναι και το βασικό μήνυμά μας. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι ε, η δέσμευση από πλευράς γονέων. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και οι γονείς αν θέλουμε να έχουμε κατάλληλη εκμάθευση, εκμάθηση την υπηρετική ηλικία και κυρίως για τα ευάλωτα παιδιά, διότι θα μπορέσουμε να έχουμε ίσως και προγράμματα για τους ε, γονείς. Ε, μία ιδέα που είναι πολύ σημαντική είναι να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη ε, κοινοτικών προγραμμάτων, να υπάρχουν ε, ευκαιρίε για τα μέλη τη κοινότητα, για την τοπική κοινότητα, να μπορούν να συναντώνται και να υποστηρίζουν ταυτόχρονα την εκμάθηση και ανάπτυξη των παιδιών τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι οι οικογένειε νιώθουν ότι μπορούν να ασχοληθούν από κοινού και να βασιστούν στο κοινό του συμφέρον για τα παιδιά. Θα υπάρχει δηλαδή προσέγγιση που θα επικεντρώνει στο παιδί με την κατάλληλη συμμετοχή και των γονέων. Πολλές φορές οι νηπιαγωγή και, τα, ε, και οι όσοι ασχολούνται με το τομέα της υγείας δεν γνωρίζουν πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες αυτοί για την ανάπτυξη των παιδιών στο μέλλον. Θα μπορούσε να υπάρχει ίσως και κατάλληλη επιμόρφωση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ε, σημειώσουμε και την συμμετοχή των ε, ε, πατέρων να μην γίνεται διάκριση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, να γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ειδικές ανάγκες και η πρόληψη, η κατάλληλη διαπίστωση αν αυτό γίνει από πρώιμη ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ε, προσεγγίσουμε τις οικογένειες και όσους ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών ε, σε νηπιακή ηλικία. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη συνένεση, προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων αυτών των προγραμμάτων. Σε πολλά κράτη-μέλη, κυρίως για τα πιο ευάλωτα παιδιά, ε, επισημαίνεται ότι οι βελτιώσεις ε, στην πρόσβαση ε, δεν είναι κατάλληλες για να βοηθήσουν τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευάλωτα και κυρίως για τα παιδιά κάτω των τριών ετών πολλές φορές υπάρχει το πρόβλημα του χαμηλού εισοδήματος και της έλλειψης παιδείας. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε λίγο και τις διεξιότητες των ανθρώπων που φροντίζουν τα μικρά παιδιά και θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι έχουν τις κατάλληλες ε, τα κατάλληλα προσόντα και θα αναγνωρίζονται αυτά ε, από το κράτος όπως πρέπει. Ε, σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε χωρισμένη την νηπιακή ηλικία σε δύο τμήμα. Υπάρχουν υπηρεσίες από 0 έως 3 ετών και από 3 έως 6. Σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται κατάλληλες ομάδες των υπηρεσιών και δημιουργούνται αρκετά προβλήματα διότι δεν γίνονται τα πάντα προς όφελος του παιδιού. Εάν λοιπόν ε, στην έκθεση αυτή ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν κατάλληλα ολοκληρωμένα συστήματα, ε, θα έχουμε κάποια πρόεδρο. Υπάρχει βέβαια η Δανία, η Σουηδία και η Φιλανδία που έχουν ανάλογα συστήματα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μάθουμε και εμεί κάποια πράγματα από αυτά. Επίση, θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα τη πρόσβαση στι υπηρεσίε αυτέ. Σε πολλά κράτη-μέλη αυτέ οι υπηρεσίε είναι αρκετά ακριβέ που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν αντέχουν οικονομικά το βάρος αυτό και υπάρχει και όλη η συζήτηση για το ποιος και ε, πότε θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να αγγίξουμε και αυτό το θέμα. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τι γίνεται με τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών και να υπάρξει κατάλληλη ανταλλαγή, διότι όπως σας είπα υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο στην ηλικία των 2 ετών μπορούν αλλά δεν υποχρεωμένα να πάνε στο σχολείο μέχρι τα 6 τους χρόνια ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο στα 5 τους και σε κάποιες περιπτώσεις και στα 4. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερος εξορθολογισμός ώστε η νηπιακή ηλικία να εξετάζεται κατά νήνων. Δεν είναι απλώς ένα επιπλέον βάρος, είναι τμήμα του συστήματος και θα πρέπει να εξετάσουμε το σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταλλάξουμε και εμπειρίες. Νομίζω επίση ότι είναι κρίμα ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και προγράμματα όπω το Κομένιο, στο οποίο επιτρέπει στου διδάσκοντε να συμμετέχουν σε συστήματα ανά την Ευρώπη, δεν ε, είναι αρκετά γνωστά και θα πρέπει ε, να ε, γνωστοποιηθούν ακόμα περισσότερο σε όσου παρέχουν υπηρεσίε εκμάθηση για τα παιδιά σε νηπιακή ηλικία. Επίση, χρειαζόμαστε και στοιχεία αυτή τη στιγμή τα στοιχεία για τα μικρά παιδιά είναι πολύ ε, ε, ελάχιστα, είναι διάσπαρτα την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχουμε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες ε, εκμάθησης νηπιακής ηλικίας και τους παιδαγωγούς στην ηλικία αυτή. Όπως σας είπα νωρίτερα, τα περισσότερα στοιχεία που έχουμε είναι από τις αγγλόφωνες χώρες και κυρίως από τις Ηνωμένε Πολιτείε και νομίζω ότι αυτό δεν είναι πολύ ε, σχετικό και περιορίζει πολύ και το πεδίο μας διότι δεν καλύπτει αυτά που αναζητούμε. Τα Ηνωμένε Πολιτείε δεν μοιάζουν σε καμία περίπτωση με καμία από τις χώρες μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ακριβώ υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα υπηρεσιών νηπιακή ηλικία, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε είναι μία ε, συγκριτική μέθοδο ανά χώρα, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να μάθουν το ένα από τα άλλα. Για παράδειγμα, ε, πολλοί γονείς και επαγγελματίε. Ε, θεωρούν ότι η κατάλληλη εκμάθηση θα πρέπει να γίνεται σε μια σχολική αίθουσα, που νομίζω ότι αυτό δεν είναι και το κατάλληλο μοντέλο. Το σκανδιναβικό μοντέλο δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο σημασία έχει το να υπάρχει και εκμάθηση και διδασκαλία εκτός αιθούσης. Ε, Επίσης θα μπορέσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσουμε και να επικαιροποιήσουμε τους στόχους μας ε, όταν θα έχει συσταθεί το σύστημα εκμάθησης νηπιακής ηλικία. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία. Συνεργαζόμαστε και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μιλήσω και με την Ουγγρική Προεδρία για το θέμα αυτό σε ε, δύο εβδομάδες περίπου, στη διάρκεια της Πράσινης εβδομάδα, και ε, συζητήσαμε πολλά και με το γραφείο της κυρίας Βασιλείου. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική δουλειά και τα τρία θεσμικά όργανα συνεργάζονται επί του θέματος και ελπίζω να υπάρχει και υποστήριξη από όλους εσάς για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Χάνιμπαλ. Να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το 2002 ήδη ασχοληθήκε με το θέμα αυτό στη Βαρκελόνη και δήλωσε ότι μέχρι το 2010 θα πρέπει να έχουν αλλάξει πολλά στον τομέα αυτό. Τι διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Σε κάποιες χώρες έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, αλλά όχι τόσο λόγω εκπαίδευσης, αλλά λόγω των ικανοτήτων των ε, μητέρων. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις ε, που τα παιδιά πηγαίνουν σε ε, σταθμούς φύλαξης. Ε, στη δική μου χώρα υπάρχουν περιθώρια μεγάλης ε, πρόοδου. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί δυστυχώς κρέμεται από πάνω μας ο πάθος του, ε, της επικρικότητας. Μπορούμε να ελπίζουμε και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υποβάλει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις τις οποίες θα υποστηρίξει το Κοινοβούλιο και θα περάσει το Συμβούλιο προκειμένου να πετύχουμε κάτι για να αναρωτηθούμε μετά από ένα-δύο χρόνια τι πετύχαμε. Και όπως είπε η κυρία Χάνιμπαλ υπάρχουν καλά παραδείγματα από χώρες από τις οποίες μπορούμε πολλά να μάθουμε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ μεταξύ άλλων στόχων ε, για το 2020 θέλουμε να περιορίσουμε το ποσοστό του 15% των ατόμων που δεν ολοκληρώνουν την σχολική εκπαίδευση σε 10%. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε γρήγορα από πρώιμη ηλικία την ε, σωστή υποστήριξη των παιδιών. Κυρίως για τα παιδιά εκείνα τα οποία δεν έχουν ε, δυνατότητες και πρόσβαση στην εκπαίδευση από το σπίτι τους όπως έχουν άλλα παιδιά. Σας ευχαριστώ για την ε, εξήγησή σας και της παρουσίασή σας, ο συνάδελφο Τσφέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το Σας ευχαριστώ. Μιλάμε για την ε, πρώτη περίοδο μαθητείας στη ζωή του παιδιού. Υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία. Όχι, όχι. Ε, η αγγλική καμπίνα δουλεύει τώρα, γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ε, εντάξει, δουλεύει. Ευχαριστώ τη συνάδελφο που ανέλαβε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπήρχε ένα κενό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και τη συγχαίρω πραγματικά για την πρωτοβουλία της αυτή. Νομίζω ότι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον εξαρτάται και από τις οικονομικές επενδύσεις και από την προσπάθεια που καταβάλουμε για να προάγουμε το μέλλον των παιδιών μας. Τα πρώτα χρόνια, όπως είπε η κυρία Χάνιμπολ, είναι τα πιο σημαντικά. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος στην ανάπτυξη του παιδιού και, στην ε, και σε ό,τι αφορά τις γνωστικές ε, λειτουργίες και σε φυσικό επίπεδο αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικά αυτά τα χρόνια. Υπήρχε λοιπόν αυτό το κενό το οποίο δεν είχαμε ε, λάβει καθόλου υπόψη μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάποιες θετικές πολιτικές, κάποιες καλές πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν καλά μοντέλα σε κάποια κράτη-μέλη και μάλιστα και κάποια από τα νέα κρατημέλη, Κάποιε από τις ανατολικές χώρες έχουν ε, καλές πρακτικές να μας προσφέρουν και να εμπνεύσουν τα παλιά κρατημέλη. Παραδείγματο χάρη η Σλοβενία και η Τσεχία είναι τέτοιε περιπτώσει. Είναι αρκετά εμπεριστατωμένη η έκθεση. Λείπουν φυσικά κατά τη γνώμη μου κάποια πράγματα παρόλα αυτά. Δεν αναφέρουμε αρκετά θέματα υγείας και διατροφής. Αλλά μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου έχουμε ακόμα χρόνο για να βελτιώσουμε το κείμενο και να κάνουμε τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Βαρκελόνης, ε, την εποχή εκείνη ούτε εμείς δεν ήμασταν σίγουροι για το ποιες ήταν οι καλές συστάσεις στον τομέα αυτό για την ε, ηλικία από 3 έως 6 χρόνια είχε γίνει η σύσταση ότι το 90% των παιδιών θα πρέπει να έχουν τέτοια νηπιακή εκπαίδευση. Αλλά σε νωρίτερη ηλικία, 0 έως 3, οι ειδικοί είχαν πει ότι το 1 τρίτο αρκεί να έχει πρόσβαση σε τέτοιε ε, υπηρεσίες. Αυτές οι στάσεις νομίζω ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν, γιατί και τα πρώτα-πρώτα χρόνια ε, είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει πολύ περισσότερα παιδιά να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποκτήσουν διατάξεις ούτως ώστε ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών να συμπεριληφθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα ήδη από την υπιακή ηλικία. Γιατί τα παιδιά αποκτούν και γνωστικές λειτουργίες ε, και άλλες ε, δεξιότητες που είναι πολύ σημαντικές και θα είναι υποφελείς και για την υπόλοιπη ζωή τους. Πρέπει να κάνουμε ακόμα πάρα πολλά σε αυτόν τον τομέα. Ακούσα ότι ετοιμάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία έκθεση και ελπίζω ότι και η δική μας έκθεση, καθώς και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ενθαρρύνουν μία μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφο Τάκουλα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Χάνιμπον για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι έκανε μια θαυμάσια προσπάθεια Άκουσα την παρουσίασή της. Νομίζω ότι ήταν πλήρης, συμπεριέλαβε όλα τα βασικά σημεία. Θα πρέπει να χτενίσουμε λίγο ακόμα το κείμενο, ούτως ώστε να δώσουμε έμφαση στα πιο σημαντικά σημεία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν οι πόροι Εδώ δεν μιλάμε για την ενέργεια. Δεν μιλάμε ούτε για τίποτα μαγικό. Μιλάμε για τους νέους και για τα παιδιά μας. Και δεν θα πρέπει να τους ξεχνάμε. Θα πρέπει να τους θυμόμαστε πιο συχνά και σε άλλες επιτροπές. Όχι μόνο στη δική μας επιτροπή, να μην μιλάμε για τους νέους μόνο στην Επιτροπή Πολιτισμού. Η συγγήτρια. Τόνισε ότι από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου συμβαίνουν σημαντικά πράγματα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που κυκλοφορούν με βάση τις οποίες τα τρία πρώτα χρόνια ή τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου το παιδί έχει μια εξαιρετικά γρήγορα, γρήγορη ανάπτυξη και στη συνέχεια απλώς επαναλαμβάνουμε ένα κύκλο ο οποίος μοιάζει με τον πρώτο αυτό κύκλο 0 έως 3 ή 0 έως 5. Να μην το ξεχνάμε αυτό, το λένε πολύ ειδικοί. Εδώ μιλάμε για τα νήπια. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι παιδιά. Θα πρέπει σε όλη αυτή την προσπάθεια να μην ξεχνάμε και την σημασία του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού και ειδικά του νηπίου. Δεν θα πρέπει να μιλάμε από την αρχή για την, τις απαιτήσει της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινα όντα και θα πρέπει να τους προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για να αναπτυχθούν. Μιλήσαμε πολύ για τις γνωστικές δεξιότητες και για άλλες δεξιότητες που αποκτά το παιδί, ήδη από τα πρώτα χρόνια. Μιλήσαμε για την άθληση, ε, για τη φυσική γενικά δραστηριότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, ούτω ώστε να επιτρέψουμε στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού να αναπτυχθεί. Χαίρομαι για την προσπάθεια που έκανε μέχρι στιγμή η συγγήτρια και είμαι πεπισμένος ότι η τελική μας έκθεση θα είναι πολύ ποιοτική. Τα προβλήματα που παραμένουν είναι να πείσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν όλες αυτές τις ιδέες και να αλλάξουν τον τρόπο δράσης τους, ώστε να προχωρήσουμε. Σημείωσα με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα παιδιά αλλά και τους γονείς, και τον πατέρα και τη μητέρα. Ε, πρέπει να υπάρχει μια καλή οικογενειακή ατμόσφαιρα, ευελιξία στην προσπάθειά μας, ασφάλεια στο πλαίσιο αυτό. Όλα αυτά τα βασικά στοιχεία πρέπει να υπάρχουν για να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για τα παιδιά. Ε, σας ευχαριστώ ακόμα κυρία Χάνιμπολ και σας συγχαίρω για τη δουλειά σας. Ε, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Χάνιμπολ για αυτή την πρωτοβουλία. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, και την εκπαίδευσή τους και η καθολική φύση αυτών των προτάσεων ε, είναι η καλύτερη προσέγγιση. Θέλω να τονίσω και το ρόλο των γονιών και το γεγονός ότι ίσως και ήδη θα πρέπει κάπως να διαπαιδαγωγηθούν. Για να... Θα πρέπει λοιπόν να διαπαιδαγωγηθούν οι ίδιοι για να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους με τη συνέχεια. Είναι σημαντικό και τι μπορούν να προσφέρουν αυτοί στα παιδιά στο σπίτι. Επίσης, ε, η έρευνα και η ανταλλαγή καλών ε, πρακτικών είναι πολύ σημαντικό. για αυτή την ηπιακή ηλικία. Ε, η σημασία λοιπόν αυτής της έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική και χαίρομαι που μπήκε στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Και εμένα με εντυπωσίασε η δουλειά που έκανε η κυρία Χάνιμπαλ και την ευχαριστώ. Διερωτώ με αν κάπου στην έκθεσή της και το ρωτάω αυτό, θα μπορούσε να λάβει υπόψη το γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ένα θέμα με τα παιδιά των μεταναστών. Υπάρχουν κάποιες τελετές αυτών των, κάποια τελετουργικά αν θέλετε αυτών των οικογενειών που δεν γίνονται σεβαστά σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αναφέρθηκε η αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος κάνει τι θέλει. Μερικές φορές όπως στην Ιταλία, ε, ακόμα και κάποιες περιφέρειες θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Κάπου λοιπόν η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη της περισσότερο αυτό το θέμα. Κάπου να το αναφέρει. Γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλές χώρες. μην ξεχνάμε ότι αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά των μεταναστών, μαθαίνουν και αυτά και γίνονται και αυτά ε, μέσα από την, μέσα της, ε, εκπαιδευτική διαδικασία Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ να σας υπενθυμίσω ότι η κυρία Χάνιμπολ το θέμα της ε, φύλαξης και της υποστήριξης των παιδιών που προέρχονται από δύσκολες ε, δύσκολα περιβάλλοντα, το έθιξε. Ίσως θα μπορούσαμε να θίξουμε και το θέμα των μεταναστών. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, στον κύριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να καλωσορίσει αυτό το σχέδιο έκθεσης, γιατί πρόκειται για έναν τομέα πολιτικής, ο οποίος ως τώρα δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή. Ιδιαίτερα τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία θίγονται στην έκθεση αυτά είναι αυτά που χρήζουν πιο πολύ εξέταση. Θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης ε, συνδύασε πολλά σημαντικά στοιχεία για την πρώτη ε, παιδική ηλικία και για την σχετική εκπαίδευση και τόνισε γιατί είναι σημαντικά τα στοιχεία αυτά και πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά κρίσιμη η εκπαίδευση αυτή στην πρώιμη νηπιακή ηλικία για τη μετέπειτα ποιότητα ζωής, αν φυσικά υπάρχει καλή οργάνωση και σωστή ποιότητα. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται πλέον εκτίματα και για την εκπαίδευση, μπορεί να αντισταθμίσει ενδεχόμενα ψυχολογικά μειονεκτήματα και μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά μεταναστών ή μειονοτήτων και να τα βοηθήσει να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό που έχουν. Όπως και να έχει, αυτή η πρώιμη ε, εκπαίδευση είναι πιο αποτελεσματική από τη μετέπειτα ε, παρέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει σύντομα μια ανακοίνωση για την ε, εκπαίδευση για την πρώιμη νηπιακή ηλικία και αναμένουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη συμπληρωματικότητα προς την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πω ότι η έκθεση της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ επίκαιρη γιατί η Ουγγρική Προεδρία έχει επιλέξει το θέμα αυτό ως ένα από τα θέματα προτεραιοτήτων της και θα συζητηθεί στα τέλη του Φεβρουαρίου. Θα υπάρξουν και σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου το Μάιο σε ό,τι αφορά για τη συνεργασία και τη σχολική εκπαίδευση το 2008 στα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και το 2000 ε, και, το πρόγραμμα, και στο πρόγραμμα για το 2020 απευθύνεται έκκληση προς τα κράτη-μέλη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συντονισμό στον τομέα αυτό. Θεωρώ ότι το σχέδιο έκθεσης αυτό αποτελεί μία υποστήριξη για αυτό το μελλοντικό μας έργο. Όπως αναφέρεται υπάρχει μεγάλο εύρος πρακτικών και παραδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ μεγάλο δυναμικό για να μάθει μία χώρα από την άλλη σε ό,τι αφορά τις πολιτικές προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτές. Άρα θέλουμε να υπάρξει τέτοια συνεργασία στο μέλλον και θα θέλαμε να υποστηρίξουμε περαιτέρω και να συνεργαστούμε περαιτέρω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάνιμπολ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Να σχολιάσω κάποια ζητήματα. Καταρχάς, εσείς κυρία Πακ μιλήσατε για τα άτομα που δεν τελειώνουν τη σχολική του εκπαίδευση. Το αναφέρομαι αυτό στην έκθεση και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο των ε, φιλοδοξιών μας. Ξέρω ότι είναι ένα στόχος της Επιτροπής μας να μειώσει δηλαδή το ποσοστό των ατόμων που δεν ολοκληρώνουν την ε, σχολική εκπαίδευση και υπάρχει πολύ μεγάλο πάρα πολλές έρευνες οι οποίες καταδεικνύουν ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση από νωρίς οι μαθητές ε, τείνουν να ολοκληρώνουν την σχολική τους εκπαίδευση. Υπάρχει λοιπόν σχετικό α, όφελος και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε πιο έντονα. Συμφωνώ. Ε, κύριε Σφέν, το θέμα της ε, κινητικότητας, μάλλον της κίνησης, της άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο θέμα της διατροφής. Πολύ καλά ζητήματα αυτά που θίγεται και πιστεύω ότι μπορούμε να το αναφέρουμε ως τροπολογίες αν το 90% ω ποσοστό των παιδιών που θέλουμε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ασφαλώ είναι πολύ καλό στόχο, Κυρία Τάκουλα, όταν ξεκίνησε αυτή η έκθεση και ξεκίνησε η ανταλλαγή απόψεων, μιλήσατε για παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα, δεν θέλουμε να... Είπατε ότι τα παιδιά πρέπει να μένουν παιδιά, φυσικά. Δεν θέλουμε να τα επιβαρύνουμε πέραν του δέοντο Δεν είναι αυτό ο σκοπό μα. Σκοπό μα είναι να είναι καλή η εκπαίδευση και η φροντίδα από τα πρώτα τους χρόνια για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά. Και φυσικά, αναφέρατε κυρία Μαρκλάκη, για το τι μπορούν να κάνουν οι γονείς στο σπίτι. Φυσικά αυτό θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουν και οι γονείς και το τονίζουμε αυτό στην έκθεση. Και θα πρέπει να υποστηριχθούν οι στο έργο του αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και περνάμε στο τελευταίο σημείο τη συζήτηση για τα παιδιά των μεταναστών. Μιλώ στην έκθεση για παιδιά από μειονεκτικέ οικογένειε. και φυσικά τα παιδιά των μεταναστών ε, μοιραία πολλές φορές ε, έχουν διπλό μειονέκτημα. Εγώ έχοντα ζήσει στο Λονδίνο μετά από την ε, επαγγελματική μου εμπειρία γιατί ήμουν και διευθύντρια στο σχολείο πρέπει να σας πω ότι είδα πολλά παιδιά που δεν ήταν ε, αγγλόφωνα. Είναι πολλές οι εθνικές μειονότητες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μου αρέσει ο όρος αυτός, αλλά περιγράφει αρκετά σωστά την κατάσταση. Και πολύ συχνά βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται πιο πολύ υποστήριξη. Χρειάζεται λοιπόν ειδική υποστήριξη για τα παιδιά των μεταναστών και φυσικά μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Όχι μόνο ωφελεί τα παιδιά και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας που αναφέρουμε στην έκθεση, αλλά δεν χρειάζονται σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μία υπόταξη αν θέλετε, ε, μεταναστών που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Άρα έχουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να αντιμετωπίσουμε τι ειδικέ ανάγκε που έχουν τα παιδιά των μεταναστών. Μου άρεσαν τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάρηκα για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού που θα χρησιμοποιηθεί. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και ανυπομονώ να ανακληρώσω, να ανακληρώσω τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τέλη Φεβρουαρίου, στις 9 μάλλον Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις σχετικές της συστάσεις στο θέμα αυτό και υποθέτω ότι η κυρία Χάνιμπαλ, η οποία έχει ήδη πολύ καλές επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τις ε, μελετήσει επισταμένως και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα προσαρμόσει και την έκθεσή της. Και αυτό φυσικά ισχύει και για όλους μας, προκειμένου να μην χρειαστεί επιπρόσθετη έκθεση για το θέμα αυτό, αλλά να είναι μοναδική η έκθεση αυτή της κυρίας Χάνιμπολ για το θέμα αυτό και να μπορέσουμε να την ψηφίσουμε έτσι. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Ευχαριστώ την κυρία Χάνιμπαλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περνάμε στο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ένα θέμα το οποίο, το οποίο πραγματικά συναντώ πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, πιο πολύ από ποτέ. Είναι πραγματικά η λέξη κλειδί, ένα κύμα αυτό το θέμα του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και τη δημιουργικότητα, Ίσως σε κάποιε περιπτώσει να το υπερεκτιμούμε το θέμα αυτό. Ελπίζω να μα προσγειώσει όμω η Μαρή Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απαντάμε σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Απελευθερώστε το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και του ψηφιακού κόσμου μοιάζει να απειλεί αυτούς τους κλάδους, αλλά να μην ξεχνάμε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και νέες σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους. Μπορεί να βελτιωθεί το δυναμικό, υπάρχει αυτή η λέξη στον τίτλο, που ακόμα δεν έχει τύχη εκμετάλλευση αυτού του κλάδου πολιτισμού και δημιουργικότητας. Το να υπάρξει μια, έτσι, ένα ευρωπαϊκό δυναμικό για να τονώσει αυτούς τους κλάδους είναι πολύ σημαντικό. Θα σας παρουσιάσω τους βασικούς ε, άξονες με συνοπτικό τρόπο. Καταρχάς, η δυτή φύση αυτών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Καταρχάς έχουν ένα οικονομικό άξονα, δίνουν θέσει απασχόλησης, προωθούν την ανάπτυξη, δημιουργούν πλούτο και υπάρχει και ένα πολιτιστικό στοιχείο, ένας πολιτιστικός άξονας που οδηγεί στην άνθηση και στην κοινωνική ένταξη των Ευρωπαίων. Εν συνεχεία, ο σημαντικό ρόλο στην προώθηση τη πολιτιστική ποικιλομορφία και τη γλωσσική ε, επικοινωνία, του πλουραλισμού, τη κοινωνική και εδαφική συνοχή, αλλά και στον εκδημοκρατισμό ε, τη πρόσβαση στον πολιτισμό και στον, στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ε, σημαντικό ρόλο επίσης, έχουν και στην οικονομία. Την ψηφιακή εποχή ε, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προώθηση της επικοινωνίας και της ε, ενημέρωσης. Πρέπει να προβληματιστούμε ε, για τις συνθήκες εργασίας, τις οικονομικές πτυχές, φορολογικές πτυχές και νομικές πτυχές στον τομέα, στο εσωτερικό αυτών των τομέων. Και επίσης, όπως είπε και η κυρία Χάνιμπολ προηγουμένως, να αναλύσουμε αυτούς τους δύο κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας όχι γενικά, αλλά να δούμε κλάδο προς κλάδο, ούτως ώστε για να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και να καταλάβουμε ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά και τα πλεονεκτήματα. Οι δράσεις που προτείνουμε ε, είναι, βασίζονται σε έξι βασικούς τομείς. Καταρχάς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλλιτεχνική εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών, να σεβαστούμε την δημιουργία, ούτω ώστε να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, τις γνώσεις ε, και την κατανόηση των τεχνών ε, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Με την ευαισθητοποίηση από την πιο νεαρή ηλικία, με προγράμματα κατάρτισης, με τη συνεργασία ε, τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών, των φοιτητών, των μαθητών των σχολείων, των επιχειρήσεων, των τεχνητών και καλλιτεχνών, καθώς και των οργανισμών χρηματοδότησης, ε, οπουδήποτε συναντούνται οι επαγγελματίες του κλάδου μέσω του πειραματισμού και της ανταλλαγής απόψεων, της βελτίωσης των δεξιοτήτων, την ευαισθητοποίηση του μεγάλου κοινού, χάρη σε συζητήσεις, σε κατάρτιση και σε μια εταιρική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η κλάδη της, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας δημιουργούν πόλους δημιουργικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που δημιουργούν μετά με τη σειρά τους ε, μια ελκυστικότητα στην περιοχή σε επίπεδο τουρισμού, οικονομικό, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση και στην προώθηση της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς της Ευρώπης. Εν συνεχεία, με την κινητικότητα και την έλξη που ασκούν. Το να προωθήσουμε την κινητικότητα των καλλιτεχνών είναι ένα τρόπο για να βοηθήσουμε τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητα για να περάσουν από το τοπικό επίπεδο στο εθνικό επίπεδο. Εν συνεχεία, δεύτερον, η διάδοση των, ε, ψηφιακών, ε, έργων ε, την ψηφιακή εποχή με τους κατάλληλους μηχανισμούς ε, και οικονομικούς, ούτως ώστε να ψηφιοποιήσουμε όσο μπορούμε το σύνολο της πολιτικής πολιτιστική κληρονομιά. Να έχουμε επίση κοινού ευρωπαϊκού κανόνε. Νομίζω τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν πρέπει να δράσουν, τόσο ώστε να προχωρήσουν τι προσπάθειέ του ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Ε, Α μιλήσουμε για την ενιαία αγορά των, του περιεχομένου την ψηφιακή εποχή. Θα πρέπει να έχουμε καινοτόμα μοντέλα και να, ε, να προσφέρουμε νέες, νέους τρόπους ε, υπηρεσιών online. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά των υπηρεσιών online να δούμε ποιοι είναι οι φορεί, να, να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα ε, και υπηρεσίε που προωθούν την ανάπτυξη και να βοηθήσουμε του Ευρωπαίου πολίτε να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, εξασφαλίζοντα την προστασία και, τον, και τη δίκαιη ανταμοιβή των δικαιούχων. Επίση, θα πρέπει να προσαρμόσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, του κανόνε που ισχύουν σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και να τους προσαρμόσουμε στην ιδιαιτερότητα του, του, του κλάδου του πολιτισμού. Να διαδώσουμε τα έργα μέσω πρωτοβουλειών με σκοπό τη βελτίωση και της μετάφρασης, του υποτιτλισμού κτλ. Επίσης, στα νέα, στη νέα γενιά προγραμμάτων media και πολιτισμού για την επόμενη περίοδο 2014-2020 συμπεριλαμβάνοντάς τα στον προγραμματισμό των κρατών μελών όσο μπορούμε περισσότερο. Ε, να δημιουργήσουμε επίση τα κράτη-μέλη ειδικά φεστιβάλ και ειδικές, ειδικά γεγονότα. Επίσης, η διαχείριση των κλάδων αυτών. Θα πρέπει να έχουμε πολυγλωσσικές πλατφόρμες ε, όπου θα, ε, θα βρίσκονται μαζί οι επαγγελματίες να, να ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες, να συνεργαστούν στα πλαίσια πιλωτικών ή κοινών προγραμμάτων, όχι σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε διασυνοριακό και υπερεθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να έχουμε πραγματικές πληροφορίες για τους νομικούς κανόνες που ισχύουν, για να δούμε τις δυνατότητε χρηματοδότησης που υπάρχουν, να υπάρχουν υπηρεσίες ε, παροχής συμβουλών για την χρηματοδότηση και διαχείριση των επιχειρήσεων επίσης. Είναι σημαντικό να καταρτήσουμε σημαντικ... Ε, κατάλληλους επαγγελματίες, ούτως ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα ε, οικονομική και άλλη των ε, προγραμμάτων, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην πίστοση ε, και να δούμε ότι οι οικονομικοί φορεί γενικά δεν γνωρίζουν τι ιδιαιτερότητε αυτού του τομέα. Φυσικά θα πρέπει να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση αυτών των κλάδων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στρατηγικέ επενδύσει υπέρ αυτών των κλάδων. Θα πρέπει η χρηματοδότηση να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των κλάδων αυτών. Θα πρέπει να έχουμε και νέα οικονομικά καινοτόμα εργαλεία, παραδείγματο χάρη τραπεζικές εγγυήσεις, κεφάλαια υψηλού κινδύνου κτλ. Επίσης, δράσεις ευαισθητοποίησης ε, στις υπάρχουσες δυνατότητες ε, χρηματοδότησης. Επίσης, τεχνική αρρωγή να μην ξεχνάμε τη σημασία που μπορούν να παίξουν τοπικές και περιφερειακές αρχές για να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνάντηση των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και των οργανισμών που μπορούν να τις χρηματοδοτήσουν. Να χρηματοδοτήσουν αυτούς τους κλάδους, να ευαισθητοποιήσουμε τους ε, χρηματοδοτικούς οργανισμούς ε, και να τους ε, γνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα αυτών των κλάδων να γνωρίσουν τη φύση τους, ότι κυρίως αποτελούνται αυτοί κλάδοι από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, να δημιουργήσουμε μικροχρηματοδότηση βραχίας διάρκησης για την προώθηση και ανάπτυξη πολιτιστικών προγραμμάτων μέσω εταιρικών σχέσεων τομέα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και γενικά όλες οι δαφικές αρχές να δικτυωθούν, ούτως ώστε να ανταλλάσσονται καλές πρακτικές και να εφαρμόζονται πιλωτικά προγράμματα διασυνοριακά και πανευρωπαϊκά, ούτω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη άμυλα στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Θα ήθελα τώρα να με βοηθήσετε με τις ιδέες σας για να τροποποιήσουμε αυτή την έκθεση, ούτω ώστε να, να απηχεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απόψεις των μελών της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Μαριτέλε. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι στην έκθεση αυτή ε, περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία τα οποία τα οποία τα συζητάμε εδώ και 18 χρόνια. Από το 1992 έγραψα, ξέρετε, την πρώτη έκθεση για το θέμα αυτό, την κατάσταση των καλλιτεχνών στην Ευρώπη και έθεσα αξιώσει τότε οι οποίε επαναλήφθησαν το 1996, το 99 σε άλλε εκθέσει και το 2000 και πριν από δύο χρόνια από άλλους συναδέλφους. Δυστυχώς λίγα έχουν συμβεί, γίνει πρόοδος και κυρίως α, μιλάμε για τη ζωή των καλλιτεχνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της κινητικότητάς τους σε ό,τι αφορά το φορολογικό καθεστώ τους ε, προκειμένου ένας καλλιτέχνης ο οποίος ε, ε, βγάζει κάποια χρήματα για τρεις μήνες και δεν βγάζει χρήματα για νέα μήνε να μην χρειάζεται να πληρώνει πέραν ποσά μόνο του τρει μήνε αυτού, αλλά να υπάρχει μια κατανομή αυτών των φορολογικών ε, ε, επιβαρύνσεων. Στην Γαλλία είναι πολύ καλό το καθεστώς για τους καλλιτέχνες και νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αναφερθούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, όχι μόνο στο πλαίσιο του κλάδου γενικότερα, αν θέλετε, αλλά να αναφερθούμε και στα άτομα που βγάζουν το ψωμί τους από το κλάδο αυτό. Ο Ιβο Μπελέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στα Ολλανδικά, μου επιτρέπετε. Γιατί είμαι συντάκτης γνωμοδότησης για την έκθεση της κυρίας Σάντσο Σμιτς από την Επιτροπή Βιομηχανίας και νομίζω ότι είναι σημαντικό το εσωτερικό της Επιτροπής Ήτρε να καταρτιστεί μία γνωμοδότηση για να καταστεί καταρχάς σαφές ότι μιλάμε για καλλιτέχνες, για πολιτισμικές πρωτοβουλίες αλλά και παράλληλα ότι μιλάμε για έναν τομέα οικονομικής σημασίας, όχι έναν ήπιο τομέα, soft τομέα, αλλά για έναν τομέα ο οποίος είναι σημαντικός για το σύνολο της οικονομίας μας. Η συμβολή του τομέα αυτού στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το 2,6% της συνολικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Πολύ σημαντικός τομέας λοιπόν. Είναι ευρύς ε, φυσικά ο ορισμός, μιλάμε ε, για τους καλλιτέχνες, τους αρχιτέκτονες, το design, ε, ο οπτικοακουστικός τομέας, όλα αυτά υπάρχονται στο σημαντικό αυτό κλάδο της οικονομίας μας στην ε, Επιτροπή Βιομηχανίας θα υπογραμμίσουμε κυρίως τις πλευρές πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτό το τονίζει και η κυρία Σάντσο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, ε, ξέρετε, συνήθως έχουν ένα και μόνο πρόβλημα, τα λεφτά. Πώς θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και να παραμείνουν βιώσιμες. Αυτό λοιπόν η πρόσβαση σε νέα χρηματοοικονομικά ε, μέσα, μέσα τα οποία ονομάζονται Angel για παράδειγμα, προκειμένου να εξοπλιστεί ο οικονομικός τομέας με νέα χρηματοδοτικά μέσα για τις μικρές εταιρείες που ασχολούνται με τα πολιτισμικά. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, ε, το θέμα του ΦΠΑ, του φορολογικού καθεστώτος των επιχειρήσεων αυτών, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Η διαφορά μεταξύ offline και online ΦΠΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει εκ νέου να το θέσουμε επιτάπητος. Ίσως δεν έχει νόημα, αλλά καλό είναι να τονίσουμε ότι ζητάμε ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις ε, παραγωγές online. Και περνάμε λοιπόν ε, σε θέματα ψηφιακής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι επίκαιρο, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θέλουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα αυτά online, ότι είναι πραγματικά αυτό πολύ κρίσιμο. Γιατί οι εταιρείες αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μόνο εφόσον γνωρίζουν ότι τα δημιουργήματά τους ε, θα προστατεύονται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ως στόχο η κυρία Κρούς. Με όλους, ξέρετε, με όσους συζητάμε από τον κλάδο μας τονίζουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Τελευταίο στοιχείο, κυρία εισηγήτρια, κυρία Πρόεδρε, είναι αυτές οι γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και του κλάδου, αλλά και μεταξύ βιομηχανίας και του τομέα της δημιουργικότητας. Είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για τη βιομηχανία, αν θέλετε, της δημιουργικότητας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επιλογή λέξεων γιατί αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει και την παραδοσιακή βιομηχανία, την βιομηχανία του χάλυβα τη βιομηχανία των αυτοκινήτων. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να υπάρξουν αυτές οι γέφυρες μεταξύ της κλασικής βιομηχανίας και της δημιουργικής βιομηχανίας και να υπάρξουν μεγαλύτερα κίνητρα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και από το κοινοβούλιο μας να δημιουργήσουμε επαφές μεταξύ του σκληροπυρηνικού, αν θέλετε, τομέα της βιομηχανίας και του κλάδου αυτού του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα. Είναι τεράστια η συμβολή της δημιουργικότητας σε ό,τι αφορά την οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των καλλιτεχνών, νομίζω ότι τα αναφέρατε τα στοιχεία τα οποία ήθελα να αναφέρω. Δεν πρόκειται να επαναληφθώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέγει η Πρόεδρο. Κύριο Κέλλη. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχά, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Έχει παρουσιάσει ε, τα θέματα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στον ε, τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, διότι πολλές φορές τους βλέπουμε ως κατακαιρματισμένους και όταν συζητάμε πραγματική πολιτική και πραγματική οικονομία, θεωρούμε ότι η κλάδη αυτή δεν είναι και τόσο σημαντική αλλά όπως είπε και ο, ο συνάδελφος Ιβο, είναι το 2,6% του ΑΕΠ και υπάρχουν πάρα πολλοί, άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ σημαντικέ θέσεις απασχόλησης. Όταν τελείωσε η συγκήτρια ήμουν πολύ ικανοποιημένη, αλλά μετά είπατε εσείς κυρία Πρόεδρε ότι η συζήτηση αυτή ε, συνεχίζεται εδώ και 18 χρόνια και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι επ' αυτού, να θέσουμε κάποιους στόχους και να πούμε ότι αυτά θέλουμε να επιτύχουμε, διότι πολλές φορές έχουμε επικρίσεις για τους πολιτικούς και την πολιτική τους και λένε ότι είναι πολλά λόγια και καθόλου πράξεις. Ήγκη και η ώρα για πράξεις λοιπόν. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω για τα θέματα των online υπηρεσιών, ε, τη διανοητική και πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό είναι ένα καθόδη ζήτημα για πολλούς συγγραφείς και καλλιτέχνες. Και είναι πολύ ε, σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται σε όλες ε, τις σε κάποιες χώρες, αναφέρατε τη Γαλλία εσείς, εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες φοροαπαλλαγές και σε άλλες χώρες για τους ε, καλλιτέχνες και τους δημιουργούς και θεωρώ ότι θα πρέπει να, θεωρήσουμε, να καθορίσουμε και κάποιους στόχους να χρησιμοποιήσουμε κάποιες ιδέες της Μαρή Τερέζ, αλλά και τη δική σου την παρατήρηση αν το θέμα αυτό διονύζεται εδώ και 18 χρόνια και κάποια θέματα δεν έχουν υλοποιηθεί, θεωρώ ότι και είναι η ώρα να δράσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να υποδείξω το εξή. Θα είχαμε κάνει κάτι αν μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι για να μην θεωρήσουν όλοι όσοι με ακούν ότι δεν κάναμε τίποτα. Όλοι το πρόβλημα είναι ότι έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γιατί για τέτοια θέματα μόνο κίνητρα μπορούμε να δίνουμε ως Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν ε, μεταφέρω αυτό το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, προς τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως είπε και η κυρία Σάντσες, θεωρώ ότι το θέμα αυτό ε, θίγει πολλά ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέρουσες πτυχές του κλάδου, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Να σας πω ότι όταν είδα την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταρχάς ήμουν κάπως, απογοητεύτηκα κάπως, γιατί μου δίνεται η εντύπωση ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα ε, περιορίζεται η θεώρηση του κλάδου αυτού ε, περιορίζεται μόνο σε θέματα οπτικοακουστικά και αυτό δεν μου αρέσει. Και πολλά άτομα τα οποία ε, δραστηριοποιούνται στον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς. Αλλά δεν θα θέλαμε να τονίζουμε έτσι αυτό, γιατί έτσι μειώνεται η αξία του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Στην πράσινη βίβλο δηλαδή, δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή στον κλάδο αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε το θέμα λοιπόν αυτό, κοιτώντα και γίνεται και στην Γερμανία. Πάντα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει κανεί να είναι προσεκτικό, γιατί ο πολιτισμό και η δημιουργικότητα και οι σχετικές, ε, τα σχετικά κίνητρα δεν θα πρέπει να οδηγούν μόνο σε ενθάρρυνση και κίνητρα στην κλασική εκπαίδευση, σε μουσεία κτλ. Να μην υπάρχει μάλλον αντίθεση σε ό,τι αφορά τους δύο τομείς αυτούς. Πρόκειται για κλάδους που είναι ξεχωριστοί ως προς τη φύση τους και η... τα κίνητρα στον τομέα του πολιτισμού δεν θα πρέπει να είναι αντίθετα σε αυτά. Είναι σημαντικό λοιπόν να το τονίσουμε αυτό και να το λάβουμε υπόψη στι διαβουλεύσεις μας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αντίφαση στους κλάδους αυτούς. Όχι. Και οι δύο κλάδοι έχουν τη δική του αξία. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται διαφορετικού τύπου κίνητρα. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό που αναφέρεται στο 5 ε, της έκθεσης της κυρίας Σάντσες ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της χρηματοδότησης και της εκπαίδευσης των καλλιτεχνών σε ό,τι αφορά τον οικονομικό κλάδο γιατί σε ό,τι αφορά θέματα δημιουργικότητας, ε, όσοι ασχολούνται με τέτοια θέματα αυτά έχουν τη δημιουργικότητα. Εκεί που έχουν προβλήματα είναι στα πρακτικά ζητήματα, στα οικονομικά ζητήματα. Δεν ξέρουν συχνά αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, τι γίνεται ε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, ε, την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Γι' αυτό λοιπόν τέτοια υποστήριξη χρειάζεται προ τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλέ πολλές ευκαιρίες συνεργασίας με διάφορα σχετικά εντρήματα και με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη προκειμένου να λάβουν ακριβώς οι καλλιτέχνες την υποστήριξη στους κλάδους εκείνους που δεν έχουν εμπειρία για θέματα τα οποία δεν διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια. Και το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση σε πίστοση. Ξέρουμε για παράδειγμα, ότι οι τράπεζες δεν είναι πάντα διατεθειμένες να χρηματοδοτούν τέτοιες μικρές δημιουργικές επιχειρήσεις, πάντα δυσκολεύονται. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ενίσχυσής μας, να μην περιοριστούμε μόνο σε θέματα μέσων, αλλά να δούμε τι γίνεται και σε θέματα δημιουργικότητας και να αναρωτηθούμε κατά πόσον μπορεί να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό και στα διευθυντικά προγράμματά μας. Ίσως να υπάρχουν και εδώ ευκαιρίες για να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Να μην περιοριστούμε στα σχετικά ασθενή, Αντίναμα να τα πω προγράμματα ενίσχυσης του πολιτισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντική, σημαντικές αυτές οι επιτυχίες για κάθε Δήμο, για κάθε κοινότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να σκεφτούμε τη συμπερίληψη των διευθυντικών προγραμμάτων. Τελευταίο ζήτημα, το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης των καλλιτεχνών. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για έναν οικονομικό τομέα, για έναν οικονομικό παράγοντα. Μιλάμε για πραγματικούς ανθρώπους. Και γνωρίζουμε ότι ιδιαίτερα σήμερα ζουν σε μια πολύ δύσκολη και επισφαλή κατάσταση. Δεν έχουν καμία ασφάλεια το θέμα των φόρων το αναφέρεται ήδη και θεωρώ ότι είναι μεγάλη η ευθύνη που μας βαρύνει για να τονίσουμε και να ζητήσουμε το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης ε, των καλλιτεχνών και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να αναπτύξουμε μέτρα, μεθόδους, προκειμένου να είναι δέουσα, αρμόζουσα αυτή η ασφάλεια των καλλιτεχνών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ε, βρίσκονται σε πολύ δυσχερή κατάσταση. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε σε κάποια σημεία να το τονίσουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Μακλέκνη. Thank you. Thank you too. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Σάνσε Σμιτ για τα όσα έκανε ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργικότητας είναι ένα πάσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουμε επενδύσεις αλλά και επανεπενδύσεις στις ε, βιομηχανίες αυτές. Και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε αυτές τις δυνατότητες, πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα, κυρίως στο διαδικτυακό κόσμο, και ε, τα προβλήματα όμως που μπορεί να προκύψουν και πώς μπορεί να επηρεάσουν τη, την εργασία τους. Κυρίως ε, ε, για το downloading και την παράνομη αυτή δραστηριότητα, να φροντίσουμε ότι ζημιώνονται για τα όσα κάνουν. Και θα πρέπει να επενδύσουμε στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να επισημάνουμε, να είμαστε βέβαιοι ότι ανταμείβονται όλοι για, την, για τον κόπο τους και, το ποιότητα, και η ποιότητα που έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαρκής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάτιμο. Ευχαριστώ. Ήθελα να υπενθυμίσω και τους καλλιτέχνες όχι από πλευράς δημιουργικότητας, αλλά τους ε, performers, αυτούς που δίνουν παραστάσεις η πρόεδρος έλεγε χθε ότι ε, είναι και εποχιακή η εργασία τους. Κάποιος μπορεί να δουλεύει τρεις μήνες και μετά να μείνει εννιά μήνες άνεργος. μένα ε, μου μιλούν πολλές φορές στην Ιταλία καλλιτέχνες, ε, ηθοποιοί, τραγουδιστές οι οποίοι έχουν μεγάλες περιόδους ε, ανεργίες οι οποίες όμως δεν αποζημιώνονται ως περίοδοι ανεργίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ίσως να χαρτογραφήσει ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη για το στοιχείο αυτό και να ζητήσει από τις κυβερνήσεις να το λαμβάνουν υπόψη και να παρέμβουν επ' αυτού, διότι είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το έθιξε και η κυρία σε αυτό το θέμα και το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Ο κύριος Μπόρους έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σάντσε Σμιτ για την έκθεση αυτή, γιατί η έκθεση αυτή ανταποκρίνεται στα ερωτήματα και στις απαιτήσει ε, πολλών ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον ε, κλάδο του πολιτισμού και που μετά τη δημοσίευση της στρατηγικής για το 2020 εκφράστηκαν πολύ αρνητικά γιατί είπαν σε αυτό το κείμενο όλα τα πολιτιστικά στοιχεία ξεχάστηκαν. Είπαν επίσης ότι δεν λάμβαμε υπόψη το ρόλο του κλάδου της, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αυτή τη στρατηγική. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση και αυτή η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων θα επιτρέψει να καλύψουμε αυτά κενά και να συμπληρώσουμε την στρατηγική του 2020. Υπάρχουν τα εξή σημαντικά θέματα εδώ. Υπάρχει καταρχάς ο οικονομικός χαρακτήρας αυτού του κλάδου, αλλά Υπάρχει και ο εκπαιδευτικός, αν θέλετε, ρόλος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτός ο παιδαγωγικός ρόλος μπορεί να είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον. Γιατί οι καλλιτέχνες μπορούν να ασχοληθούν με αυτή την πτυχή της εκπαίδευσης και μπορούμε να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μετασχηματίζονται σε καταναλωτές, σε ανθρώπους που καταναλώνουν πολιτισμό και που ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο προχωράμε, χάρη σε, αυτού του είδους την κατανάλωση. Θα υπάρξει μια πολύ σημαντική έκθεση για την ενιαία αγορά σε λίγο. Η έκθεση αυτή θα κινητοποιήσει πολλές επιτροπές και στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ιδίως σε ό,τι αφορά την ε, μεταβίβαση πολιτιστικού περιεχομένου, η, την πώληση πολιτισμικών προϊόντων στην Ευρώπη. Υπάρχει το θέμα επίσης του ΦΠΑ που τίθεται σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Ελπίζω να βρούμε λύσεις για το ΦΠΑ και για τη χρηματοδότηση της, ε, των πολιτιστικών προϊόντων. Τα ευρωπαϊκά ταμεία βοηθάνε αυτές τις δραστηριότητες. Εγώ ασχολούμαι με περιφερειακά θέματα και ασχολήθηκα λοιπόν με τέτοιες ερωτήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πολιτιστικές στον τομέα του πολιτισμού ανταγωνίζονται άλλες επιχειρήσεις. Τις συνηθισμένες θα λέγαμε επιχειρήσεις. Ο τομέας του πολιτισμού σήμερα χρειάζεται μια επιπλέον βοήθεια μέσω νέων εργαλείων. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να επενδύσουμε στον τεχνικό κλάδο και στην τεχνολογία παρά στον πολιτισμό. Θα πρέπει να έχουμε ειδικά προγράμματα για τον τομέα του πολιτισμού για να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι το ειδικό στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σκεφτεί αυτό ούτως ώστε να μην υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου του πολιτισμού και των συνήθων επιχειρήσεων. Ναι, να πω. Και η ΙΜΚΟ, η Επιτροπή ζήτησε να υποβάλουν Μάλλον, πολλέ επιτροπέ ζήτησαν να υποβάλουν γνωμοδότηση, αλλά η Επιτροπή ΙΜΚΟ δεν ζήτησε κάτι τέτοιο. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο θεωρεί ότι είναι σημαντικό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράντα. Ναι, καταρχά να ευχαριστήσω την ε, Μαρή Τερέζ για την έκθεσή της, η οποία είναι εύληπτη και δεν ξεχνάει Τίποτα. Να πω ότι σε εμά, στη χώρα μου, στον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ε, βλέπουμε μια στροφή προς τον κλάδο αυτό που δεν ήταν ε, χαρακτηριστική τα τελευταία χρόνια. Άρα ο κόσμος αναγνωρίζει την ε, σημασία του κλάδου. Και αυτό το βλέπουμε και στι δραστηριότητε του εμπορικού Μελητηρίου και αλλού. Συμφωνώ και με τη συνάδελφο και με εσά, κυρία Πακ, ότι δεν μπορούμε με τις διατάξεις της Βασιλείας 3 να καταλήξουμε σε μια χρηματοδότηση τέτοιας επιχείρησης. Θα είναι αδύνατον να πληρωθούν οι απαραίτητοι όροι. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό υπόβαθρο ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα σε κλάδους τέτοιους όπου θα πρέπει να βρούμε, θεωρώ, εξαιρέσεις από τη Βασιλεία 3. Για την εκπαίδευση των νέων, για παράδειγμα, υπάρχουν σε εμά στην Αυστρία ιδρύματα τα οποία ασχολούνται με την εκπαίδευση σε δημιουργικά θέματα των νέων αλλά και σε οικονομικά θέματα. Εμείς φυσικά έχουμε μία επικέντρωση στην αυτοκινητοβιομηχανία Άρα αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να υπάρχει ένα συνδυασμό, να τονίσετε δηλαδή και η δημιουργική πλευρά αλλά και η οικονομική πλευρά και να βρούμε χρηματοδοτικά όργανα ακόμα και για τις πιο μικρές επιχειρήσεις, αν είναι δυνατόν, προκειμένου να μπορεί να βγάζει κανείς το ψωμί του. Γιατί είμαστε ασυνεπείς Μιλάμε καταρχάς ε, ε, για ηθοποιούς, για καλλιτέχνες που έχουν μια δέσμευση, αλλά έχουν και οικονομικά προβλήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε μια κατανομή του τομέα αυτού για να μην προσωμιώνονται τα άτομα αυτά με τους... Ε, για παράδειγμα, με, άλλα άτομα που φτιάχνουν κεραμικά και όχι πως έχω κάτι με τα κεραμικά. Ευχαριστώ, κύριε Στοιάνοφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και συγχαίρω την κυρία ε, Σάντσες Σμιτ για την πολύ ενδιαφέρουσα εκθεσή της. Το θέμα αυτό είναι άκρος ευρωπαϊκό και πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Μιλάμε για την ε, πολιτιστική ανάπτυξη, τις πολιτιστικές αξίες της Ευρώπης στην έκθεση αυτή. Θέλω να μιλήσω και να εστιάσω σε δύο ιδέες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο παρελθόν, πριν από 20 χρόνια, μάλλον τα τελευταία 20 χρόνια, υπήρξαν πολλά προγράμματα για αυτούς τους δημιουργικούς κλάδους. Και εγώ ανεπλάκην προσωπικά και αντιμετώπισα τις εξής μεγάλες δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία ήταν η φορολογία. Ο κύριος Σίβο Μπέλερ αναφέρθηκε σε αυτό το πρόβλημα. Εδώ κυρίως μιλάμε για το ΦΠΑ βέβαια, που στην Ευρώπη είναι περίπου γύρω στο 20%. και αφαιρεί περίπου το 15% από οποιοδήποτε κονδύλι χρηματοδότησης έχουμε προβλέψει. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποια φορολογικά ωφέλη. Γιατί αλλιώς φόροι όπως η φορολόγηση των κερδών, θα βαραίνουν πάρα πολύ και θα επηρεάσουν πολύ αρνητικά τον κλάδο αυτό. Το δεύτερο θέμα αφορά την εξέβρεση απαραίτητων, των απαραίτητων κονδυλίων για τα οποιαδήποτε προγράμματα στους κλάδους αυτούς. Εάν τέτοιες επιχειρήσεις ζητήσουν δάνειο μέσω των τραπεζών και ανταγωνιστούν άλλες βιομηχανίες, άλλους εμπορικούς κλάδους, άλλα προγράμματα εμπορικά, θα βρεθούν σίγουρα σε δυσμενή θέση. Σε πολύ δυσμενή θέση. Θα χάσουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Γιατί οι υπόλοιποι κλάδοι, εμπορικοί και τεχνολογικοί, έχουν ε, ταχείες αποδόσεις στις επενδύσεις. Πιο ε, ταχαία κέρδη. Αντίθετα από τα κέρδη στον τομέα του πολιτισμού, στους κλάδους του πολιτισμού. Εδώ έχουμε λοιπόν πολύ πιο αργές αποδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να κάνουμε μία πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου αλλά και Εθνικών Ταμείων που θα προσφέρουν χρηματοδότηση για τέτοιου τύπου πολιτιστικά προγράμματα. Και μάλιστα θα δίνουν δάνεια άτοκα. ή χαμηλότοκα δάνεια, τα οποία θα διευκολύνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χέλικα Τρούπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Σάντσε Σμιτ για τη δουλειά που έχει κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω να κοιτάξουμε ποιο είναι ο ορισμό του κλάδου του πολιτισμού και τη δημιουργικότητα. Γιατί αφενός έχουμε στην Ευρώπη στα διάφορα κράτη-μέλη μια υφιστάμενη καθιερωμένη κουλτούρα σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό που λαμβάνει κρατικές επιδοτήσεις. Ακόμα και αν υπάρχουν εθνικές διαφορές και αφετέρου έχουμε και τον ε, τομέα του πολιτισμού ο οποίος είναι ε, ε, προσανατολισμένος στο κέρδος. Αλλά υπάρχει μια ορχήστρα για παράδειγμα η οποία ε, μπορεί να λαμβάνει κρατικές επιδοτήσεις αλλά παράλληλα πουλάει και CD. Άρα συνδυάζονται αυτά τα δύο και πρέπει να δούμε ποια είναι τα ζητήματα εκείνα, ποια είναι τα θέματα, ποια είναι η κλάδη εκείνη. Αρχιτέκτονες, για παράδειγμα, εκδότες, μουσική, μόδα, ορχήστρες. Είναι σημαντικό να έχουμε διάκριση μεταξύ των κλάδων αυτών και των κλάδων που δεν έχουν εμπορευματοποίηση Είναι σημαντικό λοιπόν να κάνουμε τη διάκριση αυτή για να μην υπονοήσουμε ότι όπου υπάρχει εμπορευματοποίηση θέλουμε να πάψει η κρατική ενίσχυση. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για πολιτισμό και δημιουργικότητα. Να μην περιοριστούμε μόνο στις κλασικές, στους κλασικούς τομείς που απολάμβουν απολαύουν κρατική ενίσχυση. Γνωρίζω την ε, γερμανική συζήτηση. Τα τελευταία 15 χρόνια το επιχείρημα είναι ότι στην, ε, στο κλάδο τη δημιουργικότητα ε, απασχολούν πιο πολλά άτομα από ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία. Αλλά και αυτό ε, έπιασε προεκπλήξεω πολλού. πολλούς. Γιατί πολλοί δεν το γνώριζαν αυτό και αυτό ήταν το πολιτικό πρόβλημα. Μιλώντα λοιπόν για την ευρωπαϊκή προσέγγιση για το κλάδο αυτό, θα πρέπει το δυναμικό του τμήματος, αυτό, του τμήματος αυτού της ε, οικονομίας να ε, προωθηθεί. Και περνώ στην πολιτική μου αξίωση τώρα. Αν αυτό όντως ε, αληθεύει, θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή συνέπεια και συμφωνία για τον εξυγχρονισμό του τομέα της οικονομίας, γιατί μιλάμε για τομέα της οικονομίας πλέον, όχι για τομέα του πολιτισμού. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική για το 2020, γιατί τι είναι το smart growth που αναφέρεται η ευθύης ανάπτυξη, όταν δεν συμπεριλαμβάνεται το τομέας αυτό, αυτός του πολιτισμού. Ένα μεγάλο τμήμα λοιπόν τη στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τέτοιε πτυχέ σε ό,τι αφορά δηλαδή, τη στρατηγική του 2020. Προ αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσει. Η κυρία Ράινα φυσικά έχει δίκιο που λέει ότι σε ό,τι αφορά την Βασιλεία 3 υπάρχουν μικρά ε, project, μικρά σχέδια τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να χρησιμοποιηθεί εδώ πέρα το μέσο των μικροπιστώσεων σε ό,τι αφορά και πάλι την πολιτική για το 2020 θα πρέπει να οριστούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χρηματοοικονομικά μας μέσα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά. Και τέλος, για να υπάρχει συνεκτικότητα στη δουλειά μας, θεωρώ ότι το όλο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητα. Όταν δεν υπάρχει προστασία των νέων προϊόντων δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική επιτυχία και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αναφορά και σε άλλα έγγραφα τα οποία έχουμε ε, καταρτήσει προ αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο, Η κυρία Χανιμπόλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω κάποια σχόλια από την κυρία Κώστα, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ διότι είναι ασθενής. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω τις παρατηρήσεις που μου διαβίβασε. Η πρώτη είναι αυτό ακριβώ που ανέφερε και η κυρία Τρούπελ. Το γεγονός ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας είναι πολύ σημαντική ε, μοχλή καινοτομίας ε, σε αρκετούς κλάδους στη Γερμανία μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους που ασχολούνται με την καλλιτεχνική βιομηχανία από την αυτοκινητοβιομηχανία. Στο Λονδίνο έχουμε περισσότερους ανθρώπους από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το ξέρω, είναι απίστευτο το στατιστικό στοιχείο. Είναι διάσπαρτη και κανένας δεν ξέρει πολλά πράγματα για αυτούς, αλλά... Ε, Παρ' όλα αυτά είναι αρκετοί. Αυτά που συμβαίνουν συνήθω στην πολιτιστική βιομηχανία είναι, ε, δεν βγαίνουν στο φως του ήλιου. Η κυρία Κώστα αναφέρθηκε σε δύο τομεί που είναι πολύ σημαντικοί. Ο τομέα της μόδας και ο τουρισμός λέει ότι οι δύο αυτοί τομεί χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό δημιουργικότητα και επιχειρηματικού πνεύματο, γεγονό που έχει πολύ σημαντικέ συνέπειε στην οικονομία και στην εθνική ανταγωνιστικότητά τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ζήτησε μεγαλύτερη κινητικότητα και υποστήριξη για του καλλιτέχνε και όσου ασχολούνται με τον τομέα του πολιτισμού, ώστε να μπορέσουν να βρουν νέε δυνατότητε απασχόληση. Και επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει επενδύσει για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και για μη κερδοσκοπικού οργανισμού, οργανισμούς, ε, παρέχοντας πόρους στον προπολογισμό και καθορίζοντα συγκεκριμένα προγράμματα ε, για τα συγκεκριμένα προγράμματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην επικεφαλή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. Good Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Αυτό που θα πρέπει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη χαιρετίζει θερμά αυτή την ε, έκθεση. Να επισημάνω σήμερα ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός σύγκλησης ε, μεταξύ των βασικών στοιχείων ε, απάντησης που λάβαμε μετά τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου το φθινόπωρο και τα όσα αναφέρει η κυρία Σάνσε Σμιτ στην έκθεσή της. Ε, συναντηθήκαμε το Δεκέμβριο. Είχαμε 350 απαντήσεις τότε στην Πράσινη Βίβλο από ένα μεγάλο φάσμα τομέων και χωρών και διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, ε, τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο και επίσης να επισημάνω ότι οι μισοί εξ όσων απάντησαν είναι ε, φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται όχι σε ευρωπαϊκό αλλά σε ε, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ε, μας ε, ικανοποιεί λοιπόν το γεγονός ότι είχαμε ανταγωνισμό σε ε, όλα τα επίπεδα. Να αναφερθώ σε αυτά τα στοιχεία σύγκληση, διότι σχετίζονται και με πολλέ παρεμβάσει των μελών. Ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο προκύπτει σαφώ από τη διαδικασία διαβούλευση είναι η σημασία τη περιφερειακή διάσταση. Πολλοί λοιπόν επεσήμαναν πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών και τι μπορούν να κάνουν σε θέματα δικτύεση, διακλάδωση και να έχουμε και κάποια φαινόμενα τα οποία περνούν από τον έναν τομέα στον άλλον, όπω αναφέραμε και σήμερα. Ε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιώσουμε ε, τις προβλέψεις μας ως προς τις ε, γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε ε, ώστε να έχουμε δυνατότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ώστε όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα να έχουν και τα δημιουργικά στοιχεία που χρειάζονται αλλά φυσικά και τις επιχειρηματικές δεξιότητες οι οποίες είναι ολαιόνα και περισσότερο απαραίτητες. Η χρηματοοικονομική στήριξη φυσικά είναι πολύ σημαντική. Δόθηκαν και πολύ σημαντικά παραδείγματα για ε, καινοτόμο χρηματοδότηση, μικροχρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πρόβλημα ε, διότι οι περισσότεροι ε, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάποιες είναι και μονοπρόσωπες επιχειρήσεις και πολλές φορές αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες για χρηματοδότηση, ιδίως ε, επειδή είναι άειλη η φύση των προσόντων τους, είναι η δημιουργικότητα και το ταλέντο τους αυτό το οποίο πρέπει να προσφέρουν. Και κάτι το οποίο προέκυψε σαφώς από τη διαβούλευση είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, οι πτυχές αυτές ε, είναι πολύ σημαντικές, ε, πάρα πολλοί έθιξαν το θέμα αυτό και θεωρούν ότι είναι κατεπήγον το να υπάρξει κάποια δράση. Και δόθηκαν και κάποια παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να προκύψουν κάποια νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε αυτό το πλαίσιο. Ως προς το τι μελιγενέστε τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας είπα και το Δεκέμβριο, είναι στη φάση της ολοκλήρωσης. Τις τελευταίες πινελιές δίνουμε στην ανάλυση από τις απαντήσεις που λάβαμε. Έχουμε ένα έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ελπίζουμε να υιοθετήσουμε πολύ σύντομα στις επόμενες εβδομάδες και Στη συνέχεια θα υπάρξει μια ανακοίνωση η οποία προβλέπεται για φέτος το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάποιες προτάσεις πολιτικής και στρατηγικής από πλευράς ε, Ευρώπης 2020, διότι οι Υπουργοί Πολιτισμού πιέζουν για το θέμα αυτό, ζητούν ε, μεγαλύτερη αναγνώριση των ε, κλάδων αυτών στο πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Υπάρχουν κάποια καλά σημάδια αν ε, δούμε την Ευρώπη 2020 και την ψηφιακή ατζέντα. Ε, υπάρχει ανάγκη να αναγνωρίσουμε ε, την παροχή περιεχομένου και τις τηλεπικοινωνίες. Το ποιος παρέχει το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό. Και για τα θέματα της καινοτομίας υπάρχει μεγάλη ανάγκη αναγνώρισης της σημασίας του τομέα της δημιουργικότητας και του πολιτισμού για τις καινοτομίες, όχι μόνο καινοτομίες από πλευράς ε, καλλιτεχνικής, αλλά και κοινωνικής. Και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται στην ανακοίνωση του φθινοπόρου που είχαμε για την εφή e e ανάπτυξη, την περιφερειακή συνεισφορά στην FEE e ανάπτυξη. Έχουμε εξειδίκευση ε, στον τομέα αυτό και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους ε, κλάδους αυτούς, διότι ορισμένες φορές είναι ε, μοναδική για κάθε περιφέρεια και επομένω θα μπορέσουν να αποτελέσουν σημείο πώληση και δυνατότητες ε, ανάπτυξης ε, σε στρατηγικές τοπικής και περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια νέα στοιχεία, ανοίγουν κάποιες νέες πόρτες και η Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και Παιδεία σκοπεύει να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και ελπίζουμε ότι η έκθεση αυτή θα μας βοηθήσει προς αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ πολύ. Η εισηγήτρια, πολύ σύντομα. Άκουσα όλες τις παρεμβάσεις. Κανένας δεν χρειάζεται να πιστεί για τη σημασία του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Με χαρά βλέπω ότι συγκλίνουμε και αγκαλιάζουμε τις ίδιες ανησυχίες που είναι η έμφαση αυτών των κλάδων ε, που έχουν και οικονομική διάσταση αλλά και δημιουργική και πολιτιστική για την απαραίτητη χρηματοδότηση τώρα θα πρέπει να καινοτομήσουμε ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης. Η μεγάλη ποικιλομορφία αυτών των επιχειρήσεων του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου α, τις οδηγεί σε εμπόδια, ειδικά σε ό,τι αφορά τον τομέα της φορολογίας. Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες λοιπόν εδώ με αυτό το θέμα. Θα πρέπει, επίσης, το γεγονός ότι τις θεωρούμε πραγματικές επιχειρήσεις και πρέπει να τις θεωρούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Η σημασία της κατάρτισης. Εδώ και 18 χρόνια μιλάμε για αυτά τα θέματα, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει ουσιαστικά. Άκουσα να γίνεται αναφορά στα διαφορετικά ευρωπαϊκά ταμεία. Ζητήσαμε από την Επιτροπή Ρέτζι, Περιφερειακής Ανάπτυξης, να εκπονήσει μία έκθεση. Από ό,τι ξέρω όμως δεν έχει κάνει τίποτα συγκεκριμένο μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι και από πλευράς ε, Ευρώπης πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά τα διαφορετικά ταμεία, τα οποία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μπορούν να βοηθήσουν αυτέ τις επιχειρήσεις, τις πολιτιστικέ και δημιουργικές. Άκουσα τις προτεραιότητες που αναφέρει η στρατηγική 2020, θα τις αναφέρω και εγώ στην εκθεσή μου, αυτές τις προτεραιότητες. Τι γίνεται με το μικρόφωνο. Θα τις αναφέρω λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες, γιατί καλό είναι να συσχετίσουμε αυτές τις επιχειρήσεις και τον έξυπνο πολιτισμό που αναφέρει αυτή η στρατηγική του 2020, που είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Ε, επίσης, η σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχει σχετική έκθεση. Θα την κοιτάξω για να εμπνευστώ και να αναφέρω τις συστάσεις που μας αφορούν από αυτή την έκθεση. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Έχετε μπροστά σας την έκθεση Μαριτερές και μπορείτε να την εξετάσετε λεπτομερώς όλοι, να καταθέσετε τις τροπολογίες που επιθυμείτε μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. 16 Μαρτίου θα ψηφίσουμε. Σημειώστε το παρακαλώ. Ευχαριστούμε τη Μαρή Τερές, να ευχαριστήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περνάμε στο 6 της ημερήσιας διάταξης για την επαλλαγή του 2009. Γενικός προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάκτη τη γνωμοτότησής μα είναι ο κύριο Μόρτον Λέκεγκαρτ. Είναι τεχνικό το ζήτημα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορούμε να κοιτάξουμε κατά πόσο δαπανήθηκαν σωστά τα χρήματα τα οποία είχαμε προβλέψει στον προπολογισμό. Κύριε Σιλακακάρτα. Ähm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να επενθυμίσω σε κάποιους συναδέλφους αν δεν θυμούνται τι ακριβώς ε, είναι το θέμα που συζητάμε, είναι μια απόφαση μέσω της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει συστάσεων του Συμβουλίου και δηλώσεων ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ουσιαστικά κλείνει το βίο της ε, διαδικασίας προπολογισμού. Εάν εξετάσουμε τη διαδικασία, το Κοινοβούλιο θα προτείνει είτε να δοθεί η απαλλαγή είτε να αναβληθεί η απαλλαγή. Αν δούμε την ετήσια έκθεση του, Ευρωπαϊκού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, νομίζω ότι θεωρείται ότι η πολιτική συνοχή είναι ο κακός παράγοντας, αλλά επειδή είχαμε ουσιαστική μείωση Εντό τη πολιτική συνοχή, το ελεγκτικό συνεδρίο και το κοινοβούλιο ε, αναγκάστηκαν να βρουν άλλο αποδιοπομπαίο τράγο. Και δυστυχώς, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να είναι ο τομέας της παιδεία και των πολιτών ε, ο αποδιοπομπαίος ε, τράγος. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και αυτό είναι και το καθήκον που έχουμε αναλάβει για φέτο. Η εκτίμηση του ελεγκτικού συνεδρίου για τον τομέα της παιδείας και των πολιτών είναι ο εξής. Οι προκαταβολές αποτελούν το 87% των, των ε, πληρωμών, ε, δεν έχουν ε, σφάλματα και το περιθώριο σφάλματος είναι κατά 2%. Αυτό λοιπόν κατά, δεν είναι ανησυχητικό. Ωστόσο, επειδή ε, στην έκθεση γίνεται ένας απλός έλεγχος των ε, ε, πληρωμών και της λήξης πληρωμών, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλο ε, ποσοστό λαθών και ο εισηγητής επέκρινε πάρα πολύ τον τομέα της παιδείας. Τι συμβαίνει τώρα. Μίλησα με τον εισηγητή και συμφωνεί μαζί μου ότι ίσως υπερέβαλαν λίγο επί του θέματος να σας εξηγήσω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ένα 24% που είναι όμως μόνο από το δείγμα για την ε, ε περάτωση των λογαριασμών και αν δούμε το συνολικό ποσό, ε, το, τις συνολικές πληρωμές, ε, έχουμε ένα περιθώριο σφάλματος μόνο 2%. Κατ' εμέ δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθούμε εκτός και αν ε, το επιθυμείτε διακαώς αν δούμε την ε, Επιτροπή μας, εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να αποδείξουμε στις άλλες Επιτροπές και το Συμβούλιο ότι τα όσα δαπανούνται για την παιδεία καλώς δαπανούνται. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ε, διατηρήσουμε τον ίδιο προπολογισμό ή να αυξήσουμε τον προπολογισμό για την παιδεία για του χρόνου. Και νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο και φυσικά δεν θα έπρεπε η παρανόηση του εισηγητή να γίνει η γενικότερη άποψη των ε, υπολείπων συναδέλφων του Κοινοβουλίου για την, ε, τον τομέα της παιδείας. Γι' αυτό λοιπόν στο σχέδιο γνωμοδότησης μου προσπαθώ να δημιουργήσω μια κάποια ισορροπία λέγοντας ότι ε, λόγω διεύρυνσης έχουμε κάποιες ε, τάσεις ε, μείωσης και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το περιθώριο σφάλματος να είναι κάτω του 2%. Νομίζω ότι αυτό είναι πάντα ένας καλός στόχος. Στο σχέδιο γνωμοδότησης αναφέρεται επίσης ότι το σύνολο των συναλλαγών στον τομέα αυτό γίνεται μέσω εθνικών υπηρεσιών διότι Ορισμένες φορές ε, θεωρείται ο κακός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στην πράξη είναι τα κράτη-μέλη και οι φορείς ε, στα κράτη-μέλη που είναι αυτοί οι οποίοι διεξάγουν το συγκεκριμένο καθήκον και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Βέβαια, να γνωρίζουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδράμει τις εθνικές υπηρεσίες και επίσης το σχέδιο γνωμοδότησης αναγνωρίζεται και ε, το γεγονό ότι χρησιμοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά μέσα για τις αιτήσει και έτσι έχουν απλουστευτεί οι διαδικασίε αιτήσεων. Επίσης, ε, θέλουμε να μειώσουμε περαιτέρω τις καθυστερημένες πληρωμές για να έχουμε έγκαιρες πληρωμές. Τώρα το χρονοδιάγραμμα. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Θα ψηφίσουμε στις 3 Μαρτίου εδώ στην Επιτροπή. Περιμένω λοιπόν τις τροπολογίες σας και θα δω κατά πόσον θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τους κοιόδης ε, συντάκτες. Εάν θεωρηθεί απαραίτητο θα το λάβω υπόψη. Σας παρακαλώ ενημερώστε με και θα γίνει και συνεδρίαση. Ε, θα ήθελα και την άποψή σας, αλλά όπως σας είπα έχω ήδη μιλήσει με τον εισηγητή και νομίζω ότι έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα υπερβάλλουμε στο σημείο αυτό και νομίζω ότι θα λήξει το θέμα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λόκεγκαρτ. Θα ήθελα να μου πείτε, εξετάσατε προσεκτικά το πού, ε, από πού προέρχεται το 2% σε ποιους τομείς, πού μπορούμε να έχουν γίνει αυτά τα λάθη, σε αυτά τα μικρά ποσά που δίδονται, που πρέπει όταν ε, κάποιο ζητά 5.000, 2.000, 10.000 ευρώ, πώς μπορούν να υπάρχουν τέτοια λάθη. Και μήπως αυτό ε, αποτελεί ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Και είναι τεχνικής φύσεως ασφαλώς να προσπαθήσω Προσπάθησα και εγώ μάλλον να το θέσω όταν ε, συνομίλησα με τον εισηγητή και μου υποσχέθηκε ότι θα μου απαντήσει εν ευθέτο χρόνο. Γιατί φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί απάντηση στο θέμα αυτό. Ελπίζω να τη λάβω για να μπορέσω να σας πω συγκεκριμένα στοιχεία. Ωραία, ευχαριστώ. Κυρία Τρούπελ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Θα μας απαντήσεις λοιπόν, θα μας υποβάλεις και κάποιες καινούργιες ιδέες για το 2%. Λίγο πολύ Είμαι σύμφωνη με την πρόταση αυτή. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω στο σημείο 5 όπου αναφέρεται ότι συστήνει νομίζω καλύτερα να πούμε αντί για recommend urges the Commission Καλή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι λίγο πιο έντονη διατύπωση. Δεν έχω όμως ε, κατ' ουσίαν κάποια αντίρρηση. Ευχαριστώ. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ο κύριος Νάουτς λέει πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι καταρχάς ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο εισηγητής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πανικοβαλόμαστε στον κλάδο μας. Υπήρξαν κάποιες παρανοήσεις, κάπως ίσως να διωγγώθηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν, ίσως και λόγω ατυχής διατύπωσης της έκθεσης. Να σας πω ότι πριν ε, δύο εβδομάδες η Επιτροπή Βασιλείου ε, παραβρέθηκε σε ακρόαση στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό εξήγησε το φαινόμενο αυτό στην Επιτροπή και ο εισηγητής τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο μας κάνει φλάγκ για τρία θετικά ε, παραδείγματα ότι έχουμε υπογράψει ε, δηλώσεις διαβίβασης με τις εθνικές αρχές ότι έχουμε ε, σχετικές συμφωνίες και το καθεξής. Νομίζω ότι ο περιορισμός, αν θέλετε, της ζημιάς έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά ασφαλώς και θα θέλαμε να συμβάλλετε και εσείς προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα της κυρίας Πακ, το που, από που προέρχεται το 2% των σφαλμάτων, λόγω της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται από το ελεγκτικό συνέδριο, ε, ένα project, ένα σπάλμα μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο ποσοστό, το συνολικό. Για παράδειγμα, ένα project για την νεολαία, μιας και τυχαίνει να δειγματοδοτήβεται, ε, μάλλον το ποσοστό σφάλματο ήταν 100% στο project αυτό, γιατί ε, ήταν μία έγκυρη η υποβολή των σχετικών στοιχείων και αυτό πλησιάζει το 1% συνολικά. Άρα αυτό ευθύνεται και μόνο για το 1% του 2% του συνολικού ποσοστού σφάλματος που έχουμε. Και να σας διευκρινίσω ότι όλα τα σφάλματα ήταν σε επίπεδο εθνικών ιδρυμάτων, όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ασφαλώς το σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να μειωθούν και να παλευτούν τα ασφάλματα αυτά. Αυτό αποτέλεσε άλλη μια παρανόηση στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Θεώρησε η Επιτροπή ότι αυτό το κεφάλαιο αποτελούσε ένα παράδειγμα της αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και τελικά από ό,τι εξηγήσαμε ήταν θέμα εθνικών ιδρυμάτων. Μία τελευταία παρατηρήση Φυσικά συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια δυνατή για να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος, αλλά θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και να προσέξουμε σε ό,τι αφορά το κόστος του ελέγχου. Το ολοβάρος του ελέγχου θα πρέπει να λεφθεί υπόψη. Είναι αρκετά καλό το σύστημα που έχουμε θέσει σε εφαρμογή να μην υπερβάλλουμε. Λοιπόν, ασφαλώς πρέπει όπου γίνεται να λάβουμε επιπρόσθετα μέτρα. Ευχαριστώ. Ναι, έχω άλλη μια ερώτηση, λέει η Αυτό το ποσοστό σφάλματος το οποίο αναφέρατε. Τι έγινε, κατάχρηση του χρήματο αυτού, είναι χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν σε λάθο σκοπό. Τι ήταν. Όχι, δεν έγινε απάτη. Ε, το πρόβλημα ήταν διοικητική φύσεω ή θέμα επιλογή. Πάλι κλείνει το μικρόφωνο της Επιτροπής. Στην περίπτωση για την οποία σας μίλησα, το πρόγραμμα ήταν τεράστιο, με πολλούς συμμετέχοντες. αλλά υπήρχαν πολλοί συμμετέχοντε, ε, υπεράριθμοι θα έλεγα. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να ήταν επιλέξιμοι, αλλά ήταν υπερβολικά πολύ άριθμοι. Δεν είναι, δεν είναι απάτη αυτή, αλλά έπρεπε να είχε εντοπιστεί το πρόβλημα. Ε, μιλάμε για τέτοιου τύπου ή και για τέτοιου τύπου σφάλματα. Για φοιτητέ τώρα, για το έρασμους επίσης, ε, και εκεί υπήρχαν ε, προβλήματα, λάθη. Παραδείγματο χάρη πόσο καιρό μένει ε, ένας φοιτητή σε ξένη χώρα, πέντε μήνες, έξι μήνες, και αν έχει επαρκείς αποδείξεις. Ε, ορισμένοι, ας πούμε, πληρώνουν για έξι, ε, πληρώνεται μάλλον κάποιος φοιτητής για έξι μήνες, αλλά δίνει αποδεικτικά στοιχεία μόνο για πέντε μήνες. Τέτοιου τύπου, ας πούμε, σφάλματα εντοπίζει το ελεγκτικό συνέδριο. Άρα αυτό το παράδειγμα δεν είναι πολύ κακό παράδειγμα. Δηλαδή, τι να σας πω, μιλάμε για εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε τα άτομα πάνω από 28. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Και εγώ αυτά τα δύο παραδείγματα ε, που άκουσα. Τα μόνα δύο μάλιστα παραδείγματα που έχω ακούσει είναι αυτά που είπατε κι εσείς. Το θέμα είναι πόσο χρήμα και πόση προσπάθεια πρέπει να δαπανίσουμε για να περιστύλουμε αυτά τα σφάλματα. Και θα αναφερθώ και σε αυτό στην έκθεση και σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Ελπίζω να μην είναι πολύ άριθμε. Είναι η 1η Φεβρουαρίου, 3 Μαρτίου θα ψηφίσουμε. Σα ευχαριστώ κύριε Λοκιγκάρτ για την ε, εργασία σα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δήλωση που έκανα. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, Youth on the Move, νεολαία σε κίνηση, ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων επαγγελματική κατάρτιση. Έχουμε κάνει ήδη μία ανταλλαγή απόψε με τον συνάδελφο Τσβέρ, ο οποίο ήταν στη Σλοβενία υπουργό ε, παιδεία στο παρελθόν. Και νομίζω ότι τώρα θα έπρεπε να παρουσιάσετε το σχέδιο έκθεσή σα. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Η πρώτη ανταλλαγή στην Επιτροπή μας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ πλούσια. Ακούστηκαν και επικρίσεις, ε, ζητήθηκαν επίσης διευκρινήσεις. Και συμφωνήσαμε για τον τρόπο λειτουργίας αυτής της εμβληματική πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι η ανταπόκριση ήταν ε, πολύ καλή. Η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών επίσης ετοίμασαν από μια γνωμοδότηση καθεμιά. Και είναι η μοναδική εμβληματική πρωτοβουλία για την οποία η δική μας Επιτροπή είναι υπεύθυνη. Δεν θα ξεχνάτε ότι αυτό είναι το τμήμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που μιλάει για την έξυπνη, σφαιρική και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι στόχοι είναι δύο. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω μεγαλύτερης κινητικότητας και δεύτερον, μια ευκολότερη μετάβαση στην αγορά εργασίας για όλους όσους έχουν ολοκληρώσει τον εκπαιδευτικό τους κύκλο. Είναι μια αμφίβια προσπάθεια, για να το πω έτσι. Εν μέρη είναι, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και εν μέρει έχει επαγγελματικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή Απασχόλησης ε, θα ασχοληθεί με την απασχόληση, με το τμήμα της απασχόλησης και εμείς με το τμήμα της παιδείας. Ίσως υπάρξουν κάποιες συγκρούσεις με την Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα τα δύο τμήματα, εκπαίδευση και απασχόληση. Τώρα, τι περιμένουμε από αυτή την πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, το θέμα είναι να μειώσουμε αυτούς που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο, να βελτιώσουμε την ε, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην ε, επαγγελματική κατάρτιση. Δεν μιλάμε μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, λοιπόν, αλλά και για την επαγγελματική κατάρτιση. Τονίστηκε αυτό πολύ σημαντικά, πολύ έντονα στην ε, πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, ε, δεν μιλάμε μόνο για την επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για την άτυπη. Και σε αυτούς τους τομείς θέλουμε να επιτύχουμε πρόοδο. Όπως θα ξέρετε, η ανώτατη εκπαίδευση είναι από τους πιο σημαντικούς τομείς αυτής της πρωτοβουλίας. Και θέλουμε η διαδικασία της ε, Μπολόνιας να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε τα πανεπιστήμια μας να γίνουν πιο σύγχρονα να γίνουν πανεπιστήμια τρίτης γενιάς. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά στην οικονομία, πιο ανοιχτά στο περιβάλλον. Και θέλουμε τα πανεπιστήμια μας να μην ε, κάνουν εκπαίδευση και έρευνα μόνο, αλλά να πουλάνε και την τεχνογνωσία τους στους οικονομικούς φορείς. Θέλουμε πανεπιστήμια που να είναι τμήμα της κοινωνικής ζωής. Κάποια δυτικά πανεπιστήμια έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά πολλά άλλα όχι. Και ελπίζω ότι η μεταρρύθμιση της Μπολόνιας θα μπορέσει να μας βοηθήσει να φτάσουμε τους Αμερικάνους και τους Ιαπωνέζους. Πολύ σημαντικό είναι η επαγγελματική κατάρτιση. Η διαδικασία της εκπαίδευσης της Κοπενχάγης είναι πολύ σημαντική εδώ. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται πολύ έντονα με την οικονομία. Ε, επίσης υπάρχει ο δομέας της απασχόλησης. Με αυτόν όμως θα ασχοληθεί η Επιτροπή Απασχόλησης. Θέλω να συνοψίσω κάποια από τα σημαντικά στοιχεία της πρώτης μας ανταλλαγής απόψεων. Η πρόεδρος μας πιστεύει όπως ξέρετε, ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν πρέπει να ανταγωνιστεί ή να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα προγράμματα. Είναι μια πρωτοβουλία που είναι συμπληρωματική στα όσα υπάρχουν ήδη. Πιστεύει ότι η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης και θα πρέπει να φτάσουμε στο στόχο του 40%, 40% των νέων μας να ολοκληρώσουν την ανώτατη εκπαίδευσή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι 40% θα έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά 40% των ανθρώπων θα είναι πάρα πολύ ε, καταρτισμένοι με πολλές δεξιότητες και θα έχουν και δεξιότητες που τις έχουν αποκτήσει και αλλού, όχι μόνο στο πανεπιστήμιο πρόεδρος μας επίσης ότι η βαθμονόμηση των πανεπιστημίων δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Καλό θα ήταν να έχουμε μια διαδικτυακή πύλη που μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητέ ε, κατά την επιλογή των, του πανεπιστημίου τους, όταν αποφασίζουν δηλαδή για το τι σπουδές θα ακολουθήσουν. Ο κύριος Λόκεγκαρντ είπε ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να συνδέονται πιο στενά με τις επιχειρήσεις πρέπει να αρθούν τα εμπόδια, είπε, μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Η κυρία Κόμερχερντ είπε ότι η διαδικασία της ε, Μπολόνιας δεν ε, οδήγησε ακόμα σε πλήρη αναγνώριση των σπουδών που έχουν ε, αποκτηθεί και γίνει σε ξένη χώρα, στο εξωτερικό. Ο κύριος Κούρια είπε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν δημοσιονομικές δαπάνες για προγράμματα όπως αυτό που αφορούν τους νέους και ότι τα πολιετή προγράμματα για τους νέους θα πρέπει να συνεχιστούν. Η κυρία Κλέρ είπε ότι δεν θα πρέπει να εστιάσουμε μόνο στην ε, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση. Δεν θα είναι εύκολο να πετύχουμε το στόχο του 40%. Τώρα, για να το πω με δύο λόγια. Να τα πω όλα αυτά με δύο λόγια. Η νεολαία σε κίνηση είναι μια πρωτοβουλία που θα πρέπει να είναι σφαιρική. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Δεν ανταγωνίζεται, δεν αντικαθιστά υπάρχοντα προγράμματα είναι μια στρατηγική συνέχισης των υπαρχόντων προγραμμάτων, αλλά επιφέρει και κάποιες βελτιώσεις αυτά και έχει και κάποια καινοτόμα στοιχεία. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η εκπαίδευση είναι ανοιχτή, συνδεδεμένη με τον κόσμο των επιχειρήσεων και με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην καλύτερη αναγνώριση των, επαγγελματικών, των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό και να δώσουμε έμφαση και στην ε, επίσημη αλλά και στην άτυπη εκπαίδευση. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση των νέων. Περισσότερα προγράμματα. Δεν θέλουμε μόνο γενικά προγράμματα. Θέλουμε προγράμματα και για φοιτητές και για μαθητές και υπολοιπόμεθα κατά πολύ των επενδύσεων που κάνει η Αμερική και η Ιαπωνία που είναι τα πρότυπά μας. Επίσης, αντί για την ε, ταξινόμηση με βαθμούς των πανεπιστημίων, θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές πληροφορίες. Επίσης, φραγμοί θα πρέπει να φύγουν για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυτό σημαίνει περισσότερα λεφτά, ε, δάνεια αλλά και υποτροφίες για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτήν την κίνηση, σε αυτήν την προσπάθεια κινητικότητας. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι γλωσσικές ικανότητες. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις μαθητείες που θα πρέπει να είναι τμήμα των προγραμμάτων κινητικότητας και θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες πηγές ε, χρηματοδότησης κινητικότητας. Θα ήθελα να τονίσω δύο δυνατότητες. Η μία αναφέρεται και στην έκθεση της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να δίνει ε, δάνεια σε φοιτητέ και υποτροφίες σε φοιτητέ. Η άλλη δυνατότητα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτεί αντιστοίχω τέτοιες προσπάθειες. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία έρχεται να ολοκληρώσει κάποια σημαντικά προγράμματα και γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ας πούμε, έχουμε ολοκληρώσει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στα πλαίσια αυτής υιοθετούνται σημαντικές αποφάσεις για την δομή του ευρωπαϊκού προπολογισμού την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα υποστηρίξουν ε, ήπιες λύσεις, ήπιες πολιτικές ε, και εκεί θα συμπεριλάβουμε την εκπαίδευση ή άλλου τύπου πολιτικές. Όλοι μπορούμε να προσφέρουμε ο καθένας τον τομέα του με σκοπό τη βελτίωση της ε, εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα γίνει μια συζήτηση για το σημείο αυτό, για το θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε για την ε, χρηματοδότηση μετά το 2013. Ο κύριος ε, Σαλβαδόρ Γερίγα Πολιέδο θα μας επισκεφτεί και ο κύριος Σόριν επίσης θα είναι εδώ και θα συζητήσουμε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές μαζί τους. Θα συζητήσουμε την διάρθρωση του νέου προϋπολογισμού και όπως θα ξέρετε, ο νέος προϋπολογισμός θα αντανακλά την μελλοντική δομή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Περιμένω λοιπόν πραγματικά με ανυπομονησία αυτή τη συζήτηση. Καταλαβαίνω το την ευθύνη που έχω αναλάβει και σας ευχαριστώ. Θέλω να συμπληρώσουμε τώρα τις ιδέες που ακούσαμε στην πρώτη ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι την πρώτη φορά που διάβασα τον τίτλο αυτό, θεώρησα ότι πρέπει το γιαστείο, γιατί δεν ε, θεωρώ ότι είναι καλή αυτή η πρωτοβουλία. Ωστόσο, έχει τεθεί επιτάπητος και θα πρέπει να την διαπραγματευτούμε σε ό,τι αφορά τους νέους ε, τομείς, τα νέα στοιχεία αυτά, αυτές τις, ε, αυτό το skills passport. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει έπαινο. Πώς θα πετύχει οποιαδήποτε πρόοδο και γιατί αυξάνουμε την γραφειοκρατία που ήδη υπάρχει. Είχε υπάρξει μια δέσμευση σε ό,τι αφορά την απλοποίηση, για παράδειγμα, των πληροφοριών, σε ό,τι αφορά την απλοποίηση ε, ανταλλαγής μεταξύ των νέων, αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Αν δεν σημειώνουμε καλή αξιολόγηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουμε, δημιουργούμε δικό μας σύστημα αξιολόγησης. Θα πρέπει να φροντίσουμε και να επικεντρωθούμε στην ποιότητα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Δεν λέγεται επίσης τίποτα για το θέμα της ισότητας των φύλων και της ε, εξισορρόπησης των πολιτικών ως προς την διάσταση των φύλων. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή δημιουργεί την εντύπωση ότι θα πρέπει κάπου να εκπαιδεύσουμε τους νέους προκειμένου κάπου να βρουν μια θέση εργασίας και δεν ε, τονίζεται ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει και τη διάσταση αυτή. Φυσικά υπάρχει και οικονομικός παράγοντας, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της ε, κλίσης, της φυσικής κλίσης του καθενός. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε για τον κάθε άνθρωπο να προσφέρουμε σε κάθε άνθρωπο δυνατότητε και μετά να προσπαθήσουμε για τους νέους. Πρόκειται για μια ιδέα η οποία δημιουργήθηκε και η οποία όμως θα πρέπει να προσαρμοστεί σημαντικά για να μπορέσει να επιβιώσει η κυρία Πακ λέει ότι θα πρέπει να δούμε τα θετικά της έκθεσης και σίγουρα θα τα ε, εφαρμόσουμε αυτά που συντάτε. Ο κύριος Κέλλη. Ε, Ευχαριστώ πολύ. there are quite a lot of positive aspects. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία με την ευρύτερα έννοια, διότι οι φοιτητέ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, που ε, ζουν στο εξωτερικό, όπως και εγώ, ε, μπόρεσα να νιώσω καλύτερα την Ευρώπη ε, και έχουν μια καλύτερη προοπτική από σε σχέση με αυτούς που δεν ταξίδεψαν ποτέ. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και αν θέλουμε να αναπτύξουμε αυτή την ιδέα της ε, μίας Ευρώπης, της περισσότερης Ευρώπης υπό την έννοια του να ανήκει κάποιος στην Ευρώπη, ε, κάτι το οποίο δεν θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό οι περισσότεροι, όπως και οι συμπολίτες μου Ιρλανδοί. Η στόχη αυτή είναι εφικτή και είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθούν. Το να μειωθεί η εγκατάλειψη του σχολείου κατά 10% είναι σημαντικό. και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, κυρίως ε, δεδομένου ότι όπω επισημάνθηκε το 35% των θέσεων απασχόλησης θα απαιτούν, θα απαιτούν ανώτατη εκπαίδευση και ε, μεγάλο ποσοστό θα απαιτεί και επαγγελματική κατάρτιση. Το να διατηρεί λοιπόν κάποιο τη θέση εργασίας του είναι εξίσου σημαντικό με το να έχει τι κατάλληλε δεξιότητες. Υπάρχουν και ένα-δύο ερωτήσει από πλευρά μου κάποιες διευκρινήσεις αυτή η ιδέα ότι κάποιος ο οποίος μόλις ε, αυτά από το πανεπιστήμιο θα του διασφαλίζουμε ε, και θέση εργασίας, ε, τι γίνεται με τους κατόχους απολυτηρίου, γυμνασίου και ηλικίου. Κάποιος ο οποίος έχει περάσει τη διρυτροβάθεια εκπαίδευση ή πάρει και μάστερ ή και διδακτορικό δίπλωμα, θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορη πρόσβαση ε, στην αγορά εργασίας, ενώ αυτοί που δεν έχουν ανώτατες σπουδέ δεν θα μπορούν να το κάνουν. Τι γίνεται όταν κάποιος έχει ήδη περάσει στη γραμμή, έχει και μάστερ και κάποιες περιπτώσεις έχει και διδακτορικό δίπλωμα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα αυτό. όσο περισσότερου ανθρώπου καταφέρουμε να πείσουμε να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό, τόσο το καλύτερο. Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε τόσους σταζιέρ που θα έχουν μια θετική εμπειρία για την Ευρώπη, θα επιστρέψουν στις χώρε τους και θα διαδώσουν την ιδέα της Ευρώπης. Υπάρχουν λοιπόν καλές ιδέες εδώ και θα πρέπει να τι προωθήσουμε. Τέλος, συμφωνώ και με τον συνάδελφο, ο οποίος είπε ότι πρέπει τουλάχιστον κάποια από τα πανεπιστήμια να εξυγχρονιστούν, να έρθουν στο σύγχρονο κόσμο. Ε, κάποιοι έχουν μια πολύ υπερβολική άποψη για την ε, ίδια τη σημασία τους και νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα πιο ευρωπαϊκό σύστημα ε, ταξινόμησης των πανεπιστημίων ώστε να είναι πιο συγχρονισμένη με τον επιχειρηματικό κόσμο και με το τι συμβαίνει στον κόσμο γενικότερα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία λοιπόν ε, καλά εδώ στην έκθεση και μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα καλύτερα αν ε, ε, προχωρήσουμε και τα θέσουμε ως στόχους για την Ευρώπη του 2020. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σβέρ, διότι με τη δουλειά του ουσιαστικά αρχίζει να μεταμορφώνει αυτό το περίεργο μόρφωμα που είχαμε στην αρχή και να το κάνει κάτι πιο απτό, πιο σαφές και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως σημείο αναφοράς όλοι μας νομίζω ότι πλέον απόκειται σε εμά ε, να συνεισφέρουμε για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και σε κάποιες από τις πτυχές ε, οι οποίες περιλαμβάνονται εδώ στο θέμα αυτό. Ε, είναι και γενικά τα σημεία που αναφέρονται, διότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις επί των οποίων ίσως στη συνέχεια να πρέπει να εμβαθύνουμε τουλάχιστον σε σημεία που θεωρούμε πιο σημαντικά. Θεωρώ ότι αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες για την ατζέντα της Ευρώπης του 2020 και θα πρέπει να εξετάσουμε την νεολαία λαμβάνοντας υπόψη και την ε, πτυχή της ε, μόρφωσης αλλά και τον ε, χώρο εργασίας. αυτό είναι απαραίτητο. Κυρίως διότι πλέον διευκρινίστηκε και ότι ε, το θέμα και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πλέον σύγχυση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τη νεολαία. Ε, μετά από τη συζήτηση λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να προκύψουν σαφώς ε, κάποια θετικά στοιχεία και να δώσουμε και κάποιες σαφείς κατευθύνσεις και στα κράτη-μέλη ε, αλλά και τα όσα πρέπει να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσουμε ένα νέο κίνητρο για τις ε, νέες γενναίες, για το σχολείο, για την ε, παιδεία, για την επαγγελματική κατάρτιση και τον κόσμο της εργασίας εν γέννη. Κύριε ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι το πρόβλημα το οποίο επίσταται για το θέμα στο οποίο έχει κάνει πάρα πολλά ο Μίλαν είναι ότι η νεολαία σε κίνηση είναι ένα εγκάρσιο θέματα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς την νεολαία και η νεολαία απασχολεί, μάλλον δραστηριοποιείται σε πολλούς κλάδους και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα θέμα το οποίο εμπίπτει νομικός πώς το αρμοδιότητα των ε, ε κρατών μελών από τη διαδικασία της Μπολόνιας και μετά είναι ίσως ε, λεπτομέρεια αυτό σε σχέση με αυτό που θα προκύψει σε ό,τι αφορά την πρόθεση δηλαδή, της νεολαίας Θα πρέπει λοιπόν να υποστηριχθούν αφενός τα κρατη σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητε τους, αλλά αφετέρου θα υπάρχει και συντονισμός. Όλοι έχουν φυσικά την ιστορία τους και την παράδοσή τους και στην ε, παιδεία και αυτό γίνεται αντιληπτό. Κάτι άλλο το οποίο θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό θα πρέπει και θεωρώ ότι εδώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε κάτι στην ε, προσφορά και στη ζήτηση, να τα κοιτάξουμε τα θέματα αυτά. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι τομεί οι οποίοι είναι πάρα πολύ δημοφιλεί για σπουδέ, αλλά τελικά δεν αξιοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα να δίνονται κάποιες κατευθύνσεις, να δούμε, να βλέπει κανείς προς ε, ποια κατεύθυνση θα πρέπει να, σπουδε, σπουδάσει. Για παράδειγμα, στην ε, ε, Αυστρία είναι πολύ ζήτητη η τομή των θετικών επιστήμων. Κι ας μην είναι όλοι ικανοί να σπουδάσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνουν πιο, πιο πολλές έρευνες. Ίσως θα μπορούσαν να έχουν και τα κρατημέλη κάποιες προτάσεις. Και να υπάρχει όμως και συντονισμός. Προκειμένου να μην ε, υπάρχουν αντιφάσεις. Ευχαριστώ πολύ, Έλα. Ε, Μπόρις, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σβέρ Έχουμε μια πολύ καλή εγκάρσια έκθεση. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον, διότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί στη στρατηγική. Γι' αυτό άλλωστε και είναι τόσο σημαντικό το σχετικό έγγραφο για την υλοποίηση και επίτευξη αυτών των τόσο σημαντικών δικτών. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τόσο φιλόδοξους στόχους αν θέλουμε να βελτιώσουμε τον αριθμό ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση κατά 10%, αν θέλουμε να μειώσουμε τα ποσοστά των ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο προώρα, αν θέλουμε να έχουμε κατάλληλους δείκτες για ε, μια συνολική σύγχρονη εκπαίδευση που θα ξεκινά από το νηπιαγωγείο, αν θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο παιδείας ε, σε ε, το επίπεδο μόρφωσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια νέα προσέγγιση. Οι νέοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να μορφωθούν κατά νύλος, ώστε να μπορούν να βρουν και θέσεις εργασία στο μέλλον. Έχω δύο σχόλια, το ανέφερε η κυρία Ράινε. Η υποχρέωση να μορφώσουμε τους νέους είναι στα χέρια των κρατών μελών μπορεί να είναι πολύ φιλόδοξα και μακροπρόθεσμα τα σχέδια, αλλά και τα κράτη-μέλη θα, θα πρέπει να είναι εξίσου φιλόδοξα στην εφαρμογή τους, σε επίπεδο εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών. Ιδάλω θα έχουμε απλώς ένα πολύ φιλόδοξο έγγραφο και τίποτα άλλο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία προσέγγιση προηγμένου συντονισμού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης, θα ήθελα να κάνω ένα πιο διεξοδικό σχόλιο. Αναφερόμαστε στην κινητικότητα των νέων, που είναι και δική μας ευθύνη για τους νέους. Και θα ήθελα να ε, επανέλθω στη συζήτηση που είχαμε για τη Λευκορωσία στο Στρασβούργο. Ε, θα πρέπει να νιώθουμε υπεύθυνοι για το νεολαία σε κίνηση. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 70% των νέων δεν έχουν ποτέ ταξιδέψει στο εξωτερικό. Αυτό ε, ισχύει για την περίπτωση της Λευκορωσίας. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να ε, εντάξουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους στο Εράσμους, να τους... Ε, σκεφτούμε και αυτούς τους νέους ανθρώπους, ε, να τους συμπεριλάβουμε στα προγράμματά μας ε, για την περίπτωση της Λευκορωσίας, για να διορθώσουμε αυτά τα ε, τόσο λανθασμένα συστήματα όπως αυτό το, της Λευκορωσίας. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο του έκθεση. Η κυρία Τρούπελ, ναι, θα ήθελα και εγώ να τονίσω την σημασία του συντονισμού με τα κρατημέλη. Το ανέφερε και η συνάδελφος και είπε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Βαρόσο παρουσίασαν αυτό το φιλόδοξο σχέδιο για τη στρατηγική του 2020, στη Γερμανία διαμορφώθηκε ε, αρνητικό κλίμα γιατί αναρωτήθηκε ο κόσμος τι κάνει και τι έρχεται και κάνει πάλι, τι έρχονται και κάνουν οι Βρυξέλλες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, προκειμένου να μην ξέρουμε ότι είναι δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά μόνο με μια κοινή προσπάθεια μεταξύ του ευρωπαϊκού οράματος και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και κάτι από τα κράτη-μέλη μπορεί να υπάρξει επιτυχία. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που τόνισαν τη σημασία του εγχειρήματο και σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία της Μπολόνια. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσει για το πώς εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο η Μπολόνια στα διάφορα κράτη-μέλη. Δυσκολεύτηκε πολύ η Γερμανία, η Σουηδία. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να σκεφτούμε αυτή τη φιλόδοξη ε, άσκηση, θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τα λάθη που κάναμε στη διαδικασία της Μπολόνια και να ενταχθούμε εξ αυτών. Ξέρουμε ότι σε κάποια κρατημέλη, όπως και στη Γερμανία, στις ε, σπουδές bachelor, τελικά ε, είναι πιο λίγοι οι φοιτητές οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό. Άρα ε, ήταν πολύ αντιπαραγωγικό το μέτρο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να κοιτάξουμε τις εμπειρίες των διάφορων χωρών για να μάθουμε από τα παθήματα του παρελθόντος και να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα για το πώς ε, πολλά ανώτατα ιδρύματα δημιουργήσαν δομές που ε, ενθαρρύνουν το να πηγαίνουν οι φοιτητέ στο εξωτερικό. Πολλά λοιπόν μπορούμε να μάθουμε ένα από τον άλλο για να μην ξεκινάμε πάντα από την αρχή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεκκάρτ, λέει πρόεδρος. Øh, så vil jeg godt have lov til at øh, melde mig. Ας πω και εγώ την άποψή μου. Διάφοροι τόνισαν ότι όλα εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να έχουμε την σωστή προσέγγιση, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο αυτή η ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και συμφωνώ με αυτό, με αυτούς που είπαν ότι θα πρέπει να ε, συνδέσουμε αυτή την πρωτοβουλία με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Αν δεν ε, συνδέσουμε αυτή την πρωτοβουλία με την ε, ανάπτυξη και με το δυναμικό ανάπτυξης αποκλείεται να βρούμε τον προπολογισμό για αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν και στο θέμα της ανάπτυξης. Θα ήθελα ο εισηγητής να ξεφύγει λίγο από την πεπατημένη, να μην, να μην κάνει μια παρήθμιση, ένα κατάλογο καλών ιδεών σε αυτή την έκθεση, ως γίνεται συνήθως. Θα πρέπει να, ενδυναμώ, να εστιάσει σε συγκεκριμένους τομείς και να μιλήσει για το συντονισμό με άλλες πολιτικές. Εγώ προτείνω να συνδέσουμε την κινητικότητα, τη συνεχή εκπαίδευση και την σχέση με τις επιχειρήσεις. Το βασικό είναι να εξασφαλίσουμε τις δεξιότητες του νέου ανθρώπους συμπεριλαμβανομένης και της κινητικότητας, ή μάλλον η μαλλον είναι ένα εργαλείο για να αποκτήσουν τις δεξιότητες. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει χάρη σε αυτή την εστίαση μεγαλύτερη, πρωτοβουλία στην, μεγαλύτερη υποστήριξη στην πρωτοβουλία. Να κάνω ένα σχόλιο, λέει η Πρόεδρος. Ε, είναι απόλυτη παρανόηση. Δεν πρόκειται για πρόγραμμα. Το νεολαία ναι, συγκίνηση αποτελεί μια έκκληση. Μια έκκληση στην οποία, η οποία θα μας ε, παροτρύνει να συνεχίσουμε τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα όπως ε, διαβίου μάθηση, η Ευρώπη, νεολαία για την Ευρώπη, προκειμένου να τα διαμορφώσουμε με καλύτερο τρόπο για το μέλλον και κυρίως να τα διασυνδέσουμε. Σήμερα έχουμε ξεχωριστούς ε, πυλώνες, Εράσμους, Κομένιους, Λεωνάρντο Θέλουμε να υπάρχει διάδραση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με την νεολαία σε κίνηση. Τις δραστηριότητε που ήδη έχουμε, τα προγράμματα που ήδη έχουμε. Όχι να δημιουργήσουμε ένα ε, καινούριο πρόγραμμα που να τα καλύπτει όλα αυτά, αλλά στις επόμενες θητείες να το διαμορφώσουμε καλύτερα και να τα δικτυώσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός της νεολαίας εκκίνησης. Ε, έτσι το κατανοούμε εμάς και έτσι μας εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να το ανταληφθούμε το πρόγραμμα αυτό. Άρα δεν ε, κάνουμε τίποτα λάθος, δεν ε, προσθέτουμε γραφειοκρατία, απλά όλα τα προγράμματα τα οποία ήδη ενισχύουμε θέλουμε να τα δεκτυώσουμε και φυσικά θέλουμε να φροντίσουμε για αυτό που είπε η κυρία Χάνιμπαλ με την πρότασή της σε ό,τι αφορά θέματα πρώιμης ε, εκπαίδευσης ή για παράδειγμα αυτά που ακούσαμε για τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια. Όλα αυτά τι τροματίζουν το ρόλο τους. Με κοιτάει ε, θυμωμένα η κυρία Μακλάρεν στα πλαίσια της επικουρικότητας. Δεν έχουμε τίποτα. Πέρα από τα προγράμματα αυτά, ασφαλώς και θα επιχειρήσουμε να ανταλλάξουμε τις βέλτιξες πρακτικές αυτό μπορούμε, να κάνουμε, τίποτα παραπάνω. Αλλά η νεολαία σε κίνηση είναι πραγματικά υπέροχο πρόγραμμα. Και ένα θέμα είναι, ε, δεν μπορούμε αφενός να λέμε νεολαία σε κίνηση και ότι κάτι παραπάνω πρέπει να κάνουμε, αλλά αφετέρου να περιορίζουμε τον προπολογισμό τα κονδύλια σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την ανατροφή. Αν θέλουμε να δώσουμε πιο πολλέ ευκαιρίε στου Ευρωπαίου νέου, αυτό θέλουμε να πετύχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, τίποτα παραπάνω. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Και αυτό που είπατε για την ισότητα των φύλων. Αλλά κοιτάξτε, μην μα έρθει μπούμεραν αυτό, γιατί στην εκπαίδευση τα αγόρια είναι αυτά τα οποία υφίστανται αρνητική διάκριση όλα τα προγράμματα παιδείας αξιοποιούνται πιο πολύ από, τους, από τις ε, κοπέλες και τις γυναίκες παρά από τους άντρες. Αυτό λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω, θέλει κανείς να κάνει κάποιο σχόλιο. Κυρία Έριξον, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής. Χαίρομαι που μπορώ και εγώ να πω δύο λόγια. Όπως ξέρετε, η νεολαία σε κίνηση είναι μια πολύ φιλόδοξη και στρατηγική ατζέντα και όπως επεσήμανε και η κυρία Πακ, δεν πρόκειται για πρόγραμμα, πρόκειται για μια στρατηγική ατζέντα που προτείνει μια σειρά από βασικές δράσεις και φυσικά τα μελλοντικά προγράμματα σε μεγάλο βαθμό θα υποστηρίξουν τους στόχους που έχουμε στη στρατηγική ατζέντα του νεολαία σε Να σας ενημερώσω και λίγο για κάποια πράγματα, διότι ε, σας είχα κάνει μια ενημέρωση στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων την τελευταία φορά. Να σας πω ότι πλέον έχουμε ε, συζητήσει την πρωτοβουλία και περνάμε στην ε, διαδικασία υλοποίησης πλέον των βασικών δράσεων και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι Έχουμε ξεκινήσει την εφαρμογή πολλών από τις ε, δράσεις που αναφέραμε στην ανακοίνωση εγκαίρως. Ε, έχουμε προχωρήσει πολύ το ΒΕΤ με την αναθεώρηση της Μπρίζ ε, το Δεκέμβριο. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα Έχουμε ε, στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας τη συζήτηση για το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την ε, ε, κινητικότητα και την παιδεία. Είμαστε στη διαδικασία ανάλυσης όλων των πολύ διαφορετικών αποτελεσμάτων που έχουμε λάβει από τις διαβουλεύσεις για τα μελλοντικά προγράμματα, για τη διαβίου το πρόγραμμα νεολαία και δράση, το Erasmus Mundus και ούτε καθεξής και αργότερα στη διάρκεια του μηνός θα δούμε και τις βασικές επιπτώσεις ε, για την ε, πρώιμη κατάληψη του σχολείου. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά επιτάγματα και θα πρέπει να τα τονίσουμε εδώ στην Επιτροπή. Τώρα, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Μία διευκρίνηση για την εγγύηση για τους νέους, Youth Guarantee. Αν κατάλαβα καλά θα πρέπει να το επιβεβαιώσω και με τους αδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Είναι μια εγγύηση που προτείνουμε στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω εμείς, πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Η ιδέα είναι μετά από το σχολείο να υπάρχει μια κάποια μορφή χρηματοδότηση για τέσσερις μήνες ε, είτε ως επίδομα ανεργίας είτε ως ε, επίδομα έναρξης ε, του επαγγελματικού βίου εάν κάποιος δεν μπορεί να βρει μια θέση απασχόλησης. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Επίσης να πω ότι υποστηρίζω και συμφωνώ με τη σημασία του καλού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών διότι πρόκειται για ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, εθνικής αρμοδιότητες. Έχουμε πολύ καλή πείρα επ' αυτού από το πλαίσιο παιδείας και κατάρτισης και τη σχετική στρατηγική. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρξε και μεγάλη πρόοδος στη διαδικασία της Μπολόνιας, με τις αδυναμίες της βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποια πολύ καλά παραδείγματα ε, του γεγονότος ότι ακόμα και αν είναι κάτι εθνική αρμοδιότητα και πάλι μπορούμε να έχουμε πολύ καλά ε, αποτελέσματα. Είμαστε στη διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής ε, της στρατηγικής της Ευρώπης του 2020 και ορισμένες φορές ε, μπορεί να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ εμφανή, αλλά υπάρχουν αποτελέσματα. Η διαδικασία μας στο EPL, η, ανταλλαγή βέλτισαν, η ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και υπουργείων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που παρακολούθησα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. So once again, Mr. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Σφαίρα, αν θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Είμαι ευγνώμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας ετοίμασε το υλικό γιατί έτσι έχουμε την ευκαιρία να ετοιμάσουμε με καλύτερους όρους την έκθεσή μας. Θα βοηθήσει επίσης και την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών και της ΕΟΚΕ. Πέρα από τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, η ίδια η έκθεση μου φαίνεται πολύ σημαντική. Υπάρχει το πρόγραμμα για τις ικανότητες, δεξιότητες και τις θέσεις απασχόλησης στα πλαίσια των 7 εμβληματικών πρωτοβουλειών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει ετοιμάσει την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί χωρίς αυτή πώς εμείς θα πείσουμε τα κράτη-μέλη για να εκμοντερνήσουν ε, τους τομείς αυτούς. Η πρωτοβουλία προτείνει κάποιες δράσεις, οι οποίες δεν είναι ρηξικέλευθες αλλά θα συμπληρώσουν όλα όσα γίνονται και από πλευράς Κομισιόν. Όπως υπόθηκε, αυτή η πρωτοβουλία νεολαία σε κίνηση δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα προγράμματα. Θέλουμε αντίθετα να τα υποστηρίξουμε αυτά, ούτω ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα, ούτω ώστε περισσότεροι νέοι να συμμετάσχουν σε αυτά. Η Κομισιόν είπε ότι σε 10 χρόνια όλοι οι νέοι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ανέφικτο. Καλό είναι να έχουμε φιλόδοξους στόχους, αλλά όχι αδύνατους. Ο κύριος Κέλλη είπε ότι οι νέοι όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και αυτό τους επιτρέπει να καταλάβουν καλύτερα άλλα πλαίσια το δικό τους. Όχι, πρόκειται για κάτι παραπάνω από αυτό ταξιδέψουν ε, στο εξωτερικό και δουλέψουν στο εξωτερικό θα καταλάβουν καλύτερα τη δική τους κουλτούρα. Οι επιπτώσεις της κινητικότητας είναι απίστευτες. Είμαι πεπισμένο ότι με, του, με την κυρία Ναντίλοβα, τη σκιώδη ηγήτριά μου, θα ασχοληθούμε με αυτή την πρωτοβουλία σαν τα δικιά μας. Και πιστεύω ότι η επόμενη συζήτηση στην Επιτροπή θα είναι ακόμα πιο επικοδομητική από τη σημερινή και την προηγούμενη. Ούτω ή άλλω, ήδη μέχρι στιγμή έχουμε λάβει πολλά χρήσιμα σχόλια, αλλά και επικρίσει. Και οι επικρίσει είναι πολύ σημαντικέ για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευχαριστώ την σκιώδη συγγήτρια για κάποιε από τι επικρίσεις λοιπόν που εξέφρασε. Σε ό,τι αφορά τώρα την ισότητα ανδρών και γυναικών. Αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι την ε, ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτό δεν αφορά όμως την ίση ε, μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Μιλάμε για κάτι παραπάνω. Υπάρχουν διαφορές ούτως ή άλλως στο βιωτικό επίπεδο με και τον ΔΕ. Υπάρχουν ε, κάποιες περιφέρειες που είναι πιο πλεονεκτικές, πιο προνομιακές από άλλες. Επομένως θα πρέπει να ε, εστιάσουμε όχι μόνο στην ποιότητα αλλά και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Hope... Ωραία, ευχαριστώ Μίλαν. Καλή τύχη. Ελπίζω το κείμενο να είναι καλό και να εμπνευστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το κείμενό σας. Ευχαριστώ πολύ δοσιάλους, άλλους, όλους. Τώρα, συνάδελφοι, έχω μία πρόταση. Αν συμφωνείτε να αρχίσουμε να μιλάμε για το βραβείο Λουξ. Γιατί έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Μπορώ να αρχίσω να μιλάω γι' αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι το βραβείο Λουξ γνώρισε μεγάλη επιτυχία φέτος, όχι μόνο στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στις διάφορες πόλεις και στις διάφορες χώρες μας. Κάποιες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου σε πρωτεύουσε έκαναν προσπάθειες από πέρσι να προβληθούν οι ταινίε και να τα παρουσιάσουν ως, και να ακολουθήσουν μάλλον και συζητήσεις μετά την προβολή των ταινιών είναι εξαιρετικό το πάνελ για τις επόμενες ταινίε και το πάνελ αυτό το ενισχύσαμε κατά τρία άτομα και θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα στη συνεδρίαση των συντονιστών. Να προσθέσω δύο στοιχεία. Το βραβείο αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο βραβείο για ταινίε. Πρόκειται για ένα βραβείο που ε, συμβάλλει στην ε, διάθεση της ταινία αυτής και πρόκειται για ένα βραβείο το οποίο έχει ένα περιεχόμενο με ευρωπαϊκό υπόβαθρο. Αφορά είτε ένα πρόβλημα το οποίο εφίσταται και το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε ή κάτι που μας απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο, κάτι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Φέτος συζητήσαμε με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και συμφωνήσαμε τα εξή στις 8 και 9 Μαΐου, Μαΐου τις ημέρες της Ευρώπης στις διάφορες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιάσουμε την ταινία Fremde». Θα γίνουν προβολές σε όλες τις ε, πρωτεύουσες με τους εκάστοτε υπότιτλους στην γλώσσα της ε, χώρας Κατά δεύτερον, φέτος, όταν θα πρέπει, όταν θα κληθούμε να αξιολογήσουμε τις ταινίε που θα δούμε, τα... τις τρεις ταινίε που θα μας παρουσιαστούν, και πάλι θα τις προβάλλουμε σε τις προβάλλουμε ε, στις ε, χώρες μέλη και θα δημιουργηθεί, θα διοργανωθεί ένα φεστιβάλ όπου θα προβληθούν τρεις αυτές ταινίες, το φεστιβάλ Lux. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση. Θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και θα μπορέσουμε όλοι να συμμετάσχουμε. Χάρηκα πάρα πολύ ότι ήταν πραγματικά πολύ, πιο πολύ, οι πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι σημαντικό να γίνεται αφήγηση των ε, ιστοριών μας, των ευρωπαϊκών ιστοριών μας, γιατί είναι μέρος της ευρωπαϊκής παράδοσης οι ταινίε. Άρα θα πρέπει να αφιερώσουμε όλα τα μέσα για να το διασφαλίσουμε αυτό για το, με το βραβείο Λουξ ξέρετε, έχει γίνει πολύ ευρέως ε, διαδεδομένο. Ξέρετε, καθιερωθήκαμε και στην Βενετία, γιατί πλέον προβάλλονται ταινίε του βραβείου Λουξ και για πρώτη φορά ε, παρουσιαστήκαμε στις Κάνες, στο Βερολίνο. Στις Κάνες είχαμε μια ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη στην ευρωπαϊκή πολιτική των μέσων και ήρθαμε σε επαφή με τους δημιουργούς ε, των ταινιών και ανοίγουμε έτσι πόρτες οι οποίες ήταν προηγουμένως κλειστές προς εμάς. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι πέρσι στη Βενετία, όπου για πρώτη φορά προβλήθηκαν οι ταινίε, διοργανώθηκε το εξή. Η κυρία Κώστα ήταν εκεί και ο κύριος Κουρία. Κάναμε λοιπόν το εξή στα πλαίσια του βραβείου Λουξ από τις 27 χώρες καλέσαμε ένα νέο ε, από κάθε χώρα, 27 λοιπόν νέους οι οποίοι ενδιαφέρονταν για ταινίε. Δεν μπορώ να σας πω πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τα 27 αυτά νεαρά άτομα. Είδαν και οι 27 μαζί τις ταινίε αυτές. Είδανε όλες τις ταινίε, όχι μόνο τις δικές μας, ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το ευρωπαϊκό κλίμα που δημιουργήθηκε και όλα αυτά χάρη στο βραβείο Λουξ. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες να συμμετέχουμε σε τέτοιες προβολές και στις μετέπειτα συζητήσεις. Άρα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση προς τους συναδέλφους. Τι μπορείτε να κάνετε τώρα, πέρα από την 9η Μαΐου, που είναι μία ημέρα για όλους, μπορείτε να δείτε την ταινία Fremde αλλά και τις δύο άλλες ταινίες, οι οποίες ε, διατίθενται σε μία-δυο γλώσσες, όχι σε όλες τις γλώσσες. Μπορείτε να τις ε, δανειστείτε και να διοργανώσετε μία εκδήλωση στην εκλογική σας περιφέρεια. Το έκανα με διάφορες ταινίε. Πάντα θα βρείτε ένα κινηματογράφο για πιο Καλλιτεχνικέ ταινίε, ο οποίο θα είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί μαζί σας και να διοργανώσει μετά μία συζήτηση. Σας διαβεβαιώ ότι με τον τρόπο αυτό έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Έχουμε τη γραμματεία του Λουξ στην Γενική Διεύθυνση επικοινωνία. Πελτιέ είναι ο υπεύθυνο, ονομάζεται ο υπεύθυνο. Και η Μαριζέλα, μια Ιταλίδα η οποία οι οποίοι είναι ειδικοί για θέματα βραβείου Λουξ. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί τους, να τους ρωτήσετε πώς μπορείτε να διοργανώσετε την προβολή και τι χρειάζεστε. Έχετε λοιπόν κάθε ευκαιρία να βρεθείτε στο επίκεντρο της περιφερειάς σας και να συζητήσετε τα θέματα που αφορούν τους πολίτες. πρέπει πραγματικά να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες που έχετε. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να ε, ξυπνήσει το ενδιαφέρον των νέων για την Ευρώπη. Αλλά μέσα από τις ταινίε μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, γιατί πρόκειται για ένα μέσο το οποίο ελκύει τους νέους. Θα θέλαμε λοιπόν οι ταινίε αυτές να γίνονται γνωστές, να συζητιούνται και με τον τρόπο αυτό να ανοίξει ο δρόμος προς την καρδιά των πολιτών της περιφερειάς σας. Αυτά λοιπόν ήθελα να τα πω και αύριο, αλλά μιας και σήμερα είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ, το ανέφερα σήμερα. Ελπίζω λοιπόν να λάβετε το μήνυμα που σας ε, απεύθυνθα, απεύθυνα. Ε, θα, έχουμε, θα σας διαβιβάσω και ένα σημείωμα στα αγγλικά και στα γαλλικά γραπτά προκειμένου να το συζητήσετε και με τους υπάλληλους συναδέλφους σας που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή μας και σε άλλες επιτροπές φυσικά θα αναφερθεί αυτή η δυνατότητα. Αυτά λοιπόν και το βραβείο Λουξ ως Επιτροπή ε, Πολιτισμού είπαμε ότι θα διοργανωθεί ε, ακρόαση πριν το βραβείο Λουξ με εκπροσώπους υψηλού επίπεδου του τομέα της ε, παραγωγής ταινιών, όπως και άλλα έτη, θα έρθουν να συζητήσουν, να συζητήσουμε. Αλλά αυτό δεν θα προέλθει από το δικό μας προϋπολογισμό, γιατί τον έχουμε εξετλήσει με άλλες ακροάσεις. Αν έχετε ερωτήσεις, να τις ακούσω, αλλιώς ε, θα σας δώσω το έγγραφο στα αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα είστε εξίσου ενθουσιασμένοι κι εσείς και όπως και εγώ. Τα ευχαριστώ και λύεται η συνεδρίαση για σήμερα. Σε λίγο ακολουθεί συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ και γεια σας.